Well, this is now four minutes late. I'm happy that we are three colleagues in the room. I am going to go. Έχουμε τρεις συναδέλφους στην ε, αίθουσα. Θα σας πω τα των συντονιστών που μόλις ολοκληρώθηκαν για την ε, ε, η μερίσια διάταξη του Μαρτίου, οι αναφορές για τα βουλγαρικά σχολεία και έξι αναφορές Επίσης τα ιατρικά προϊόντα στην Ανδαλουσία, τι διακρίσει κατά των παιδιών και όλα αυτά θα προσθεθούν στην ημερήσια διάταξη του Απριλίου. Για τις εκθέσει και τι γνωμοδοτήσει, οι συντονιστέ αποφάσισαν ότι η ετήσια έκθεση του διαμεσολαβητή θα την αναλάβει το EFTD. Ε, έκθεση, η ετήσια έκθεση των αναφορών και της ειδική έκθεσης έχουν αναβληθεί για το Μάρτιο. Επίσης, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια γνωμοδότηση για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της ΛΥΜΠΕ για τα ελάχιστα πρότυπα για τις μειονότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο εισηγητής θα αποφασιστεί το Μάρτιο. Τέλος, μπορεί να καταθέσουμε, αν το επιθυμούμε, ε, ε, τροπολογίες για τις ε, πιλωτικές δράσεις ε, και τον προϋπολογισμό του διαμεσολαβητή, αλλά αποφασίσαμε να τα αφήσουμε ανοιχτό προς το παρόν. Αποφασίσαμε να μην γνωμοδοτήσουμε για την απαλλαγή του 2017. Όσον αφορά τις αμφισβητούμενες συστάσεις, εγκρίθηκαν όπως είχα προτείνει, με κάποιες εξαιρέσεις πιο συγκεκριμένα η 0998 και η 147, 148 και 149 που θα παραμείνουν ανοιχτές και θα υπάρχει συνέχεια. Η 0999 θα κλείσει. Όλες οι ε, αναφορές για την Καταλωνία θεωρήθηκαν μη παραδεκτές. Όσον αφορά ε, την 563, ε, 1363 και 166, αυτές έκλεισαν και όλες οι υπόλοιπες αναφορές παραμένουν ανοιχτές και θα υπάρχει συνέχεια. Όσον αφορά τις διερευνητικές αποστολές και τις ακροάσεις, οι συντονιστές αποφάσισαν ότι η επίσκεψη στην Αμόχωστο για τις 7 και 8 Μαΐου θα αποφασιστεί ε, μέσω γραπτής διαδικασίας ε, για το κατά πόσον θα γίνει, αν θα ε, αναβληθεί για άλλη ημερομηνία κλπ. Όσον αφορά την ακρόαση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες ε, που προβλέπεται για το Μάρτιο ε, και αυτό θα περατωθεί ε, μέσω γραπτής διαδικασίας για το πρόγραμμα μέσω συναδέλφων. Το δεύτερο εξάμεινο του 2018 οι ομάδες θα υποβάλουν τα για διερευνητικές αποστολές και ακροάσεις μέχρι τις 6 Μαρτίου. Τώρα, για τη συνέχεια της αναφοράς 1088 για τη ΦΑΤΚΑ αποφασίστηκε από τους συντονιστές να υποβάλουμε προφορικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο με ψήφισμα το οποίο θα ε, κατατεθεί στην Ολομέλεια του Ιουλίου του 2018. Επίσης θα υποβάλουμε και ε, πιθανά θέματα για διοργάνωση διακοινοβουλευτικής ε, συνεδρίασης με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Η προθεσμία είναι και πάλι η 6η Μαρτίου. Επιπλέον, οι συντονιστές αποφάσισαν να καταθέσουν προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ε, το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε για τις ε, ευρωεκλογέ του 2019. Μετά έδωσα μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση για το Brexit και ε, το σχετικό σχέδιο ψηφίσματος, ε, το οποίο θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Μαρτίου για τι μελλοντικέ σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένου Βασιλείου. Επίση, ενημέρωσα για την κατάσταση ε, για την δικτυακή πύλη της ΠΕΤΗ υπήρχε μια γραπτή αναφορά για το ψήφισμα για τον Brexit. Οι συντονιστές μπορεί να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Προθεσμία Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 3 η ώρα. Μετά συζητήσαμε τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος ε, του διαμεσολαβητή, αποφασίσαμε να αναβληθεί για κάποια επόμενη συνεδρίαση και ε, στη συνέχεια οι συντονιστές ε, έλαβαν γνώση κάποιων θεμάτων προς ενημέρωση και είχαμε και μια παρουσίαση από την Άγγελα για την επίσκεψη στη Λίμα, στο Περού. Αυτά λοιπόν. Τώρα, προχωράμε στην διερευνητική αποστολή στον Τάραντα και ε, χαίρομαι που βλέπω και κάποιους ε, από τον Τάραντα εδώ στην αίθουσα. Ε, η επίσκεψη έγινε τον Ιούλιο, όπως γνωρίζετε. Εγώ ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Ήταν μαζί μας η Άγχελα Βαλίνα και ο κύριος Τερικάμπρας. Και επίσης είχαμε και δύο εξοφίκιο μέλη, τον κύριο Κοτσολίνο. Καλωσορίσατε και πάλι στην Επιτροπή μας και την Ελεονορέβη. Η αποστολή ε, πήγε στα ε, εργοστάσια και έκανε μια ε, αξιολόγηση του τι ακριβώς συνέβη. Είδαμε την κατάσταση όσον αφορά τη ρήπανση και τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και των περίοικων, καθώς επίσης και μελλοντικών κινδύνων που μπορεί να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή μια πολύ όμορφη περιοχή, την περιοχή του Τάραντα. Επίσης ε, συναντήσαμε τους αναφερόμενους καθώς επίσης και ενδιαφερομένους για να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα πώς έχει κατάσταση στο Τάραντα. Υπάρχει μια διεξοδικότατη έκθεση της διερευνητικής επίσκεψης, ε, αναφέρει όλες τις συζητήσεις και όλες τις παρατηρήσεις που κάναμε κατά την επίσκεψή μας και θα πρέπει να επισημάνω ότι η αντιπροσωπεία είδε ότι οι συνθήκες είναι ακραίες και ε, Επίσης είδε και τι συνέπειες υπάρχουν ε, με τις προηγούμενες ή και τις ε, παρούσες ε, διαδικασίες, εργοστασιακές διαδικασίες ή το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαδικασίες και βλέπουμε επίσης ότι οι άνθρωποι υποφέρουν, υπάρχει σοβαρός αντίκτυπος λόγω του αέρα που αναπνέουν, τη δυσοσμία και τη ρήπανση που ε, αφορά την καθημερινή τους ζωή και σε μέρες που υπάρχει αέρας ε, είναι ακόμα και μέσα στα σπίτια τους. Ε, σε γραπτή απάντηση σε ένα ερώτημα του Κοινοβουλίου για το εργοστάσιο ΙΒΑ, ο Επίτροπος Βέλα είπε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Ξεκινήθηκε μια διαδικασία παραβάση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2010 του 75 για τις βιομηχανικές εκπομπές και της εκτελεστικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τον καθορισμό των καλύτερων ε, δυνατών τεχνικών για τον ε, χάλιβα και το σίδηρο. Αλλά επίσης αναφέρθηκε ότι Ακόμα και αν υπάρχουν ε, διαθέσιμες, μάλλον, και αν δεν υπάρχουν πιο διαθέσιμες συνθήκες, μπορεί να βελτιωθεί η διαδικασία παραγωγής. Και αυτό φυσικά μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Ε, γενικά διαπιστώσαμε ότι δεν είναι και πολύ εύκολη η λύση. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις για τον Τάραντα. Καταρχάς θα πρέπει να ε, ληφθούν αποφάσεις και να υπάρχει επιμερισμό των αρμοδιοτήτων για τρία αναπτυξιακά μοντέλα, περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, χωρίς ε, να ε, υπόκεινται τα δύο πρώτα στοιχεία στο τρίτο και επίσης μπορούμε να αντιλήσουμε και διδάγματα από το παρελθόν. Ε, η Επιτροπή νομίζω ότι πρέπει ε, να παρακολουθήσει τι συμβαίνει στο εργοστάσιο Ήλβα και στην περιοχή του Τάραντα Αιγέννη. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συμμετείχαν και είναι παρόντες εδώ στην αίθουσα και έχουμε και μια επισκέπτηρα από τον Τάραντα. η απορρίπανση του περιβάλλοντος ε, σημαίνει ότι θα είναι πιο ασφαλής η ζωή μας και αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Λοιπόν, να δώσω πρώτα το λόγο στα μέλη. Ο, κύριο Τερι, ο κύριος Τερι δεν είναι εδώ, αλλά η Άγχελα είναι εδώ. Θέλεις να προσθέσεις κάτι? Ευχαριστώ, Σεσίλια. Όχι, τα εξήγησε πάρα πολύ ωραία. Συμμετείχα και εγώ πράγματι στην αντιπροσωπή αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο αλλά και τη Γραμματεία για το έργο τους γιατί πραγματικά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η αποστολή. Θετικά αξιολογώ ε, και την έκθεση προφανώς και επίσης το γεγονός ότι λάβατε υπόψη ε, τις προτάσεις μας είναι η έκθεση πάρα πολύ εμπεριστατωμένη, λεπτομερής, ε, έκθεση πεπραγμένων πραγματικά. Θέλω να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες που έκαναν την αναφορά αυτή και μας εξήγησαν πώς έχει η κατάσταση. Είχαμε συναντήσεις και συναντριάσεις μαζί τους επί τόπου, γιατί ήταν σημαντικό να το συζητήσουμε και μαζί τους και να μοιραστούμε τις ανησυχίες τους. Και θέλω να τονίσω ότι είναι κατεπήγον το θέμα και επιτακτική ανάγκη να πληρούνται όλες οι προαπαιτήσεις ε, για την ε, έγκριση και την αδειοδότηση. Υπάρχει κίνδυνος ε, από τη ρήπανση στις κατοικημένες περιοχές και τις όμορες. Πολύ θετική η έκθεση και ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα να πω κάτι που ήθελα να πω. Θα ότι οι πολίτες συστηματικά αποκλείονται από την πρόσβαση σε ενημέρωση για την επέκταση των εργοστασίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Πιέρο από τη Γραμματεία για την προετοιμασία. Πάρα πολύ καλή επίσκεψη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σε ευχαριστούμε που ήρθες και εσύ και με την, τα υπόλοιπα μέλη της Γραμματείας φυσικά. Έχετε εργαστεί πολύ σκληρά. Εγώ φταίω που δεν το ανέφερα στην αρχή. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ πολύ ε, και εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την πρόεδρο της αντιπροσωπείας ε, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε όλη αυτή την επίσκεψη. Και Πραγματικά ε, είμαι ευγνώμων για το πώς ε, διεξήχθη το ταξίδι. Ευχαριστούμε πολύ και για όλα τα άλλα και για την τεχνική υποστήριξη στον Τάραντο. Είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε αντιμετώπιοι με πολλά προβλήματα, προεριβαλλοντικά, θέματα υγιεινής, ε, ε, όλα αυτά έχουν σχέση με την οικονομία της περιοχής, ε, με, τα γενικότερα προβλήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι δημιουργούνται προβλήματα αναπνοής ε, και για τα μικρά παιδιά. Οι ασθένειες αυτές συνδέονται με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να ακούσουμε και εκ μέρους ε, των ε, αντιπροσωπιών και εκ μέρους των φορέων της περιοχής ε, ότι έχουν προκληθεί σημαντικά προβλήματα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο το θίξαμε. Οι υγειονομικές αρχές, αυτό είναι κάτι άλλο επί του οποίου θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Οι υγειονομικές αρχές μας είπαν ότι ακόμα και αν υπήρχε πλήρη σεβασμό των προδιαγραφών, κάτι που δεν ισχύει σήμερα, ο υγειονομικός ο κίνδυνος για την υγεία ε, θα ήταν πάρα πολύ ψηλός. Κατά την άποψή μας λοιπόν ε, υπάρχει ολιγορία. Ολιγορία εκ μέρους της ε, ΕΝΗ. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, παράμετροι και αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει κανείς ε, να έχει κατά ότι πάρα πολλά πράγματα δεν λέγονται, δεν ανακοινώνονται στους πολίτες και από την Άννη και από άλλους φορείς σχετικά με την ρήπανση που έχει προκληθεί σήμερα από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Είναι λοιπόν κατά κάποιον τρόπο ε, σαφές ε, ότι υπάρχει εδώ αποτυχία των ε, διαφόρων κυβερνήσεων για την προστασία της υγείας αλλά και για την οικονομία του ταράντου παρότι έχουν δαπανηθεί πάρα πολλοί πόροι και έχει δοθεί και οικονομική βοήθεια. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή για την οποία συζητάμε σήμερα καθιστά σαφές ότι τελικά δεν πρόκειται για την εφαρμογή των βέλτιστων τεχνικών, ούτε πρόκειται για το ότι πρέπει να αλλάξει η διαχείριση. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι πρέπει να καταργηθεί ένα πεπαλαιωμένο, απαρχαιωμένο μοντέλο να ταχθούμε υπέρ μιας, ενός εξυγχρονισμού, μιας ανανέωσης που θα ε, είναι προς όφελος όλης της περιοχής και θα δώσει χώρο και φωνή ε, σε εκείνους τους πολίτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν νέες προτάσεις, να αναπτύξουν δραστηριότητες, ε, γιατί είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε, να έρθουμε σε επαφή μαζί τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας. Ε, υπάρχει το εργοστάσιο στην Ήλβα ε, και Είχαμε και την ευκαιρία να ασχοληθούμε με αυτό. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογηθούν. Η Επιτροπή ε, πρέπει να εξακολουθήσει να παρακολουθεί εκ του ε, αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα. Ο κύριος Κοτσολίνο θέλει το λόγο. Ήθελα απλώς ε, να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουμε Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το έργο σας, ε, ιδιαίτερα τα όσα έκανε το προσωπικό της Επιτροπής μας. Ε, νομίζω ότι η έκθεση αντανακλά επακριβώς ε, όλα εκείνα τα οποία διαπιστώσαμε, αναφέρει τις επισκέψεις μας και τις συναντήσεις μας, γνωρίζοντας ότι πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Κανείς από εμά δεν έχει το μαγικό ραβδάκι για να επιλύσει τα προβλήματα. Ελπίζω, θα δούμε τώρα, έχει και εκλογέ ε, στην Ιταλία, αν ε, ε, υπάρχουν νέα πολιτικά κινήματα ή εμείς τα πολιτικά κόμματα καταφέρουμε να λύσουμε το πρόβλημα του Τάραντα σε λίγες ώρες ή μερικές εβδομάδες, εμείς θα είμαστε ευτυχείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε, θα δεχτεί όλα αυτά τα θέματα. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε με τη σοβαρότητα που εργαζόμαστε. Πιστεύω ότι στην έκθεση που μας παραδώσατε έχει κάποιες υπερβολές που θα πρέπει να τις διορθώσουμε, αλλά σίγουρα το θέμα θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και να επαγρυπνούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, διότι του τάραντα δεν εξαντλείται σε μια επίσκεψη. Ε, υπάρχει και το ε, πρόβλημα της απόσταση μεταξύ αυτού που κάνουμε. Η επίσκεψη έγινε τον Ιούλιο, ε, τώρα έχουμε την έκθεση. Εν τω μεταξύ συνέβησαν πάμπολα πράγματα και θα συμβούν και άλλα μέχρι τις 19 Μαρτίου που θα υποβάλουμε τροπολογίες, τις 24 Απριλίου που θα εγκρίνουμε την έκθεση και επομένως θα πρέπει να παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά όλο το θέμα, ε, βήμα-βήμα αν θέλετε, τα όσα συμβαίνουν στον Τάραντα, να επαγρυπνούμε και γνωρίζοντας ότι ίσως μπορεί να πρέπει να αφήσουμε και παρακαταθήκη στο επόμενο κοινοβούλιο να φροντίσει να ε, παρακολουθεί και να επαληθεύει. Εγώ συμφωνώ απολύτως ε, και να υπάρχει και μια ε, αναβίωση των σχέσεων με την κοινή γνώμη και τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Διάλογος με την πολιτεία, με τις ε, τοπικές αρχές, μεταξύ θεσμικών οργάνωτων, γνωρίζοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τον Τάραντα. Αυτή τη στιγμή συζητάμε την υπόθεση της έδρας ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και ξέρουμε ότι ακόμα και μεταξύ θεσμικών οργάνων, μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου δεν γίνεται ανταλλαγή στοιχείων και εγγράφων. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα σε μια υπόθεση σαν τον Τάραντα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικά λοιπόν ε, αυτό που κάνουμε, διότι μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερη προβολή. Εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες για την έκθεση, αλλά νομίζω ότι το πνεύμα συνεργασία είναι το σωστό πνεύμα πρέπει να είμαστε αδιάλακτοι, διότι τα προβλήματα του Τάραντα πρέπει να αντιμετωπιστούν και πρέπει να δοθεί μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο σέρνουμε πίσω μας ε, ιστορικά. Ευχαριστώ πολύ. Η Ρόζα Νταμάτεχ, το λόγο. Πρόεδρε, και εγώ θέλω να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ την Λεωνόρα, γιατί η επίσκεψη ήταν ε, πάρα πολύ ε, καλή. Ακούσαμε όλους τους επιχειρηματίες, τα συνδικάτα, τους ε, πολίτες ε, που πρότειναν ουσιαστικές εναλλακτικές λύσεις. Το, από το 2014 έχουμε πάει δύο φορές στον Τάραντο για να δούμε από κοντά τη μόλυνση, τη ρήπανση αυτή που υπάρχει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήγε στον Τάραντο, στην δική μου την πόλη, για να δει τι μπορεί να γίνει. Χάρη λοιπόν των πολιτών μπορέσαμε μπορέσαμε να έχουμε ε, την αναφορά. Ευχαριστούμε τις ε, οργανώσεις. Ε, εμείς πλέον έχουμε μια ξεκάθαρη θέση όσον αφορά τα οικονομικά προβλήματα, τα προβλήματα υγείας των Τάραντο και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν οι πηγές ρήπανσης, ξεκινώντας από την Ήλβα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα μετατροπής που ε, το είναι αυτό. Ε, βεβαίως, ε, από την άλλη, ξέρουμε ότι συνεχίζονται εργασίες στην Ήλβα και σε άλλες ε, πηγές ρήπανσης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν επενδύσεις για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στην κυκλική οικονομία, στον τουρισμό, στην γεωργία. Ένα δισεκατομμύριο. Ε, μιλάμε τώρα για πραγματικό μάρκετινγκ στις ανώσιμες πηγές ενέργειας. Αν ταπανηθεί ένα δις έχουμε 13.000 θέσεις απασχόλησης. Ε, τον Ιούλιο η Επιτροπή Αναφορών έκανε αυτή την επίσκεψη αμέσως μετά την επίσκεψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και ε, στην Ήλβα θελήσαμε ε, να επισκεφτούμε τη μονάδα. Σήμερα λοιπόν πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που να αφορά την ΕΝΗ. Υπάρχει μόνο ε, μια προοπτική και γίνεται λόγος για υπεράρθμους εργαζόμενους. Αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Οι ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα της Σίλβα θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται για μια πηγή ρήπανσης. Υπάρχουν κίνδυνοι από την παραγωγή της Ένη η οποία μεταξύ άλλων ε, γνωρίζει ότι πράγματι προκαλεί αυτό το πρόβλημα και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και χρόνια ε, έχει ε, δρομολογήσει μία διαδικασία παραβάση αλλά δεν έχει το θάρρος να τιμωρήσει την Ιταλία. Όμως ε, 6.000 κάτοικοι βρίσκονται σε κίνδυνο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή θεωρώ ότι θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη το ότι υπάρχουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι όμως εργάζονται ε, κινδυνεύοντας και από το 60 δεν γίνεται τίποτα άλλο. Ε, έχουν διπλασιαστεί και οι νεκροί στο νεκροταφείο. Τώρα πια η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Δεν υπάρχουν καν θέσεις στο νεκροταφείο και γι' αυτό ε, θα πρέπει να ζητήσουμε και να μας συγχωρήσει και ο Θεός. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μαχτά. Ε, και καλωσορίσατε στην Επιτροπή Αναφορών. Επανέρχομαι, Πρόεδρε. Και ποτέ δεν έφυγα ακριβώς, πραγματικά. Ε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ενημερωτικά να πω δύο λόγια μόνο. Φαντάζομαι ότι οι Ιταλοί συνάδελφοι το έχουν. Και εγώ για άλλους λόγους ε, προέρχομαι ε, από μια τέτοια κατάσταση. Ε, ξέρετε ότι η ArcelorMittal έκανε μια πρόταση εξαγοράς και τώρα η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει σε βάθο ε, για να δει αν τηρήθηκαν όλοι οι εμπορικοί κανόνες κτλ. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτό που έμαθα πρόσφατα είναι ότι στην Ήλβα ε, το διάταγμα εκμετάλλευση θεωρήθηκε παράνομο από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ιταλίας κατόπιν καταγγελίας του Δημάρχου του Τάραντα και του Περιφερειάρχη της Απολίας. Δηλαδή, ό,τι η έκβαση και να έχουν οι Ιταλικές εκλογές θα τους αφαιρέσουν την άδεια για τη μονάδα στην Ήλβα. Ε, ακριβώς επειδή δεν ε, γίνεται σεβαστή η νομοθεσία για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Αυτή την ενημέρωση έχω πρόσφατη, πιο απο από δύο-τρεις μέρες. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να ακούσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε τον κύριο Μάρκο Γκάσπαρινέτη. Έχετε το λόγο. Θα σας ευχαριστώ πολύ που μου προσφέρετε αυτή τη δυνατότητα και θερμά συγχαρητήρια που αναλάβατε αυτή την πρωτοβουλία και αυτή την επίσκεψη επιτόπου. Στον Τάραντο, και εγώ πήγα στον Τάραντο, για τους ίδιους λόγους ε, πριν από κάποιους ε, μήνες ε, και είχαμε και εμείς εκεί μια επιτόπια επίσκεψη. Βέβαια η δικιά σας είναι πολύ πιο πρόσφατη και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Πρόκειται για το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να αναφέρω κάποια στοιχεία αυτά που θα πω είναι στοιχεία. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένα νέο διάταγμα που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση στις 29 Σεπτεμβρίου και ε, τώρα πλέον έχει εγκριθεί το νέο περιβαλλοντικό σχέδιο. Ε, το σχέδιο αυτό θα συμπεριληφθεί, θα εξαστεί όταν θα κατατεθεί η διαδικασία επί παραβάση. Ήθελα να σε ενημερώσω για, αυτή, για αυτό το διάταγμα, γιατί κατανοώ την απογοήτευση των ε, βουλευτών που νιώθουν ότι κοιμόμαστε. Κάθε άλλο, θέλω να απογραμμίσω ότι εμείς ελέγχουμε πολύ σοβαρά την καταστροφή της ΕΛΒΑ, της μονάδας αυτής, καταστροφή είναι και το λέω ξεκάθαρα, με τρεις διαδικασίες. Πρώτον διαδικασία ε, κρατικών επιδομάτων, αυτή έκλεισε το 2017 και ήταν επιτυχημένη με την έννοια ότι ζητήσαμε από την ε, Ιταλική κυβέρνηση ε, πριν χορηγήσει κρατικά επιδόματα να εφαρμόσει την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Και αυτό κατέληξε σε ζημιά ενός δις ε, του προηγούμενου διοκτήτη και οι ε, προϋποθέσεις που ορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι πρώτα εφαρμόζεται η αρχή ορυπαίνων ε, πληρώνει και μετά τα χρήματα και μετά ε, χρησιμοποιούνται, καταφεύγει κανείς τα χρήματα του φορολογούμενου. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο, όχι μόνο η Επιτροπή, γιατί αυτή η αρχή ορυπαίνων πληρώνει βρίσκεται παγιωμένη στις συνθήκες. Το δεύτερον, η διαδικασία επί παραβάση. Πολύ σωστά αναφέρθηκε από κάποιους ευρωβουλευτές. Εξακολουθεί να κρεμεί, αναθεωρείται συνεχώς ε, με βάση το νέο περιβαλλοντικό βιομηχανικό ε, πρόγραμμα που κατέθεσε Άσελορ Μετάλ. Θα περιμένουμε τις ε, αναφορές από τη Γενική Διεύθυνση Ξαγοράς. Ε, περιμένουν και αυτοί τα σχέδια της Ακομετάλ. Ε, αυτή η έρευνα θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Και έτσι λοιπόν θα μπορέσω να ενημερώσω το Κοινοβούλιο για πορίσματα στα οποία θα καταλήξουμε πριν από την δική σας την έκθεση. Δηλαδή τελικά αν υπάρξει αγοραστής και νέο περιβαλλοντικό σχέδιο και νέο διάταγμα, αυτά θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας πριν αποφασίσουμε αν θα πάμε στο δικαστήριο ή όχι, γιατί θα έχουν προκύψει νέα στοιχεία. Ε, να πω ε, και το 1,1 που κατέβαλε η οικογένεια Ρίβα ε, και το 1,2 δις ευρώ από την Άρσελο Μετάλ αν τελικά εγκριθεί η εξαγορά από την αρμόδια γενική διεύθυνση που δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, τότε ε, τα κονδύλια που θα υπάρχουν θα είναι σημαντικά. Ε, ίσως να πιστεύουμε ότι δεν αρκούν γιατί έχει, ε, υπάρχει ρήπανση και στην περιβάλλουσα περιοχή σε μία ακτίνα 20 χιλιόμετρων μπορεί κανείς ε, να ασχοληθεί με κτηνοτροφία. Αυτό λοιπόν είναι ε, μία μεγάλη καταστροφή. Αυτό το αναγνωρίζει και Arsenal Metal την προηγούμενη εβδομάδα ε, ε, εξετάστηκε το θέμα και Arsenal μετά μπορούσε να εκφράσει τις δικές της τις αντιρρήσεις γιατί μπορούν να υπάρξουν αντιρρήσεις και από εκείνη. Όλα αυτά λοιπόν ακόμα εκκρεμούν και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Αλλά μπορείτε να είσαστε σίγουροι ότι εμείς θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα λειτουργήσουμε σε απόλυτη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κασπαρινέτη. Αυτά που μας είπατε τώρα είναι πολύ σαφέστερα από οτιδήποτε έχει πει στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταστροφή στην Ήλβα, όπως το χαρακτηρίσατε κι εσείς. Πρωτοφανές είναι. Και επίσης χαίρομαι που η διερευνητική μας αποστολή και η έκθεση μας μπορεί να βοηθήσει. Και αν όταν αποφασίσει αν θα προσφύγει στο δικαστήριο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς θα προτιμούσαμε να προσφεύγατε φυσικά. Οπότε είναι πάρα πολύ αγαστή η συνεργασία μας και η απάντησή σας. Σε ευχαριστώ πολύ για τη σαφήνεια και τα ξεκάθαρα λόγια σας. Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Για τη σύσταση, για αυτό το τμήμα του κειμένου, 19 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι. Η δε ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 24 του μηνός Απριλίου. Τελειώσαμε με αυτή την αναφορά. Θα ήθελα να πω στους αδέλφους και στην Ελεονόρα και στον κύριο Κοτσολίνο και σε άλλους ότι έχω κάποιες πολύ ωραίες αστείες φωτογραφίες με όλες αυτές τις στολές που φοράμε και τα κράνη. Αν θέλετε σας ενδιαφέρει να δείτε τις φωτογραφίες στο τηλέφωνο μου, έχουμε μεγάλη πλάκα. Ωραία προχωρούμε στην ε, αναφορά 378 ε, σχετικά με το πεδίο βολής στην περιοχή Μπαρδένας Ρεάλες ε, στην αυτόνομη περιφέρεια της Ναβάρα. Απουσιάζει ο Νοφέρον, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρίσταται. Η κυρία Σαμαρέλη, παρακαλώ. Floor to you. Okay, thank you. Um, Ευχαριστώ. Λοιπόν, Διαμαρτύρεται ο αναφέρον για τις δραστηριότητες άσκηση εκεί στο πεδίο βολής, ε, στην ε, Παρδένες Ρεάλες, στην Ναβάρα. Είναι προστατευόμενη περιοχή, είναι ε, φυσικό πάρκο και ρεζέρβα βιοσφαίρας προστατευόμενη περιοχή από την UNESCO, από την Οδηγία Habitat και τους οικοτόπους κλπ. Η προστασία λοιπόν αυτού του χώρου ως φυσικού πάρκου, δρυμού, από την UNESCO κτλ. Όλα αυτά είναι εκτός του πεδίου αρμοδιότητων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι βάσει της οδηγίας Habitat για τους οικοτόπους ε, στατεύεται η περιοχή και μάλιστα συμπίπτει με άλλες δύο περιοχές που έχουν ε, χαρακτηριστεί ιδιαίτερη αξίας προστασίας με την οδηγία για ε, τα πτηνά. Αλλά δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη κατά στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Παρ' όλα αυτά, για τα, κράτη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να αποφεύγουν να ενοχλούν τα είδη τα οποία είναι προστατευόμενα και να καταστρέφουν το περιβάλλον και τη φύση. Θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ενώ επιτρέπεται η στρατιωτική δραστηριότητα να διασφαλίζονται και να διαφυλάσσονται οι οικότοποι και τα είδη της πανίδας και της χλωρίδας. Έχουν εκφραστεί όμως ανησυχίες από πολλούς και από πολλές επανειλημμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επιπλέον πληροφόρηση από τις Ισπανικές Αρχές σχετικά με το κατά πόσο συμμορφούνται οι δραστηριότητε του πεδίου βολής με τις υποχρεώσεις που έχουν από τις οδηγίες Habitat και ε, τις ε, οδηγίες για τα πτηνά. Η απάντηση λοιπόν των Ισπανικών Αρχών ε, μας λέει ότι από το 1951 λειτουργεί εκεί το πεδίο βολής έχουν γίνει μελέτες για να εκτιμήσουν πώς επηρεάζει το περιβάλλον το πεδίο βολή και δεν έχουν καταλήξει σε καμία επιδείνωση του περιβάλλοντος ή των προστατευόμενων. Ούτε ενοχλούνται ιδιαίτερα τα διάφορα είδη, τα ζωικά από τι δραστηριότητε του πεδίου βολή και τις βολές που κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλύσει και τα κείμενα που έλαβε στα πλαίσια αυτή τη αναφορά, συμπεριλαμβανόμένη και τη έκθεση. επιστημονική έκθεση είναι αυτή, για την παρακολούθηση του ε, πληθυσμού των ε, πτηνών στον Πάρδενας ρεάλισ. Είναι το 2014 η έκθεση αυτή και έχει εντοπίσει ότι έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές, η παρουσία ε, ορισμένων ειδών ε, πτηνών ε, ως προς τη χρονική τους παρουσία εκεί λόγω των βολών. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα με την αναπαραγωγή των πτηνών. Η μελέτη καταλήγει ότι θα πρέπει περαιτέρω να διερευνηθούν αυτές οι στρατιωτικές και δραστηριότητες στους πληθυσμούς των πτηνών ε, θα πρέπει να υπάρχει και ένα σωστό σχεδιασμό όσο και έλεγχος ε, των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και των βολών έτσι ώστε να μην υπάρχουν ε, αρνητικές επιπτώσει στα πουλιά και όπως και σε άλλα είδη προστατευόμενα που βρίσκονται στι περιοχές αυτές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι το Δεκέμβριο αυτή η περιοχή εντάχθηκε και στο άρθρο 4.4 της οδηγίας Habitat και εγκρίθηκε ένα σχέδιο διαχείρισης. Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο αυτό το 2018 και από ό,τι φαίνεται η έκθεση του 2014 λήφθη υπόψη για τις συστάσεις αυτές και το επιχειρησιακό σχέδιο, σχέδιο διαχείρισης μάλλον για εκπονηθεί νέα μελέτη ως προς τον αντίκτυπο των στρατιωτικών δραστηριοτήτων στα πτηνά που προστατεύονται και συνδέονται με την οδηγία Habitat. Βάσει αυτής της πληροφόρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, είναι σε θέση να διαπιστώσει παραβίαση περιβαλλοντικού δικαίου, ούτε έχουμε καμία ένδειξη ότι οι βολές εκεί επηρεάζουν ε, αρνητικά Ε, τις περιοχές Natura 2000 ως προς Βελινεκές και τις ε, δραστηριότητες. Στις 20 Φεβρουαρίου είχαμε επιπλέον πληροφόρηση αλλά δεν ήρθαν νέα στοιχεία που ε, μπορεί να μας οδηγήσουν στο να αλλάξουν την απόφασή μας. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και να πω επίσης ότι είχαμε καλέσει και τις αρχές της Ναβάρας αλλά αρνήθηκαν να έρθουν. Ο λόγος τώρα στους συναδέλφους, η Ρώσα Ισταρά κούτ. πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, λίγο πολύ θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα προσπαθήσω να κάνω μια παρέμβαση για να ρίξουμε και λίγο φως στην υπόθεση. Πρόκειται για ένα πεδίο βολής σε μια περιοχή που είναι ε, περιοχή ε, κοινοτικού ενδιαφέροντος και ε, το πεδίο βολής όμως υπάρχει και από το 1951. Ε, έχουν περάσει όλοι οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι και σε καμία περίπτωση, ε, σε καμία οδηγία δεν υπήρχε κάποια παραβίαση και δεν υπήρχε κάτι το οποίο να ήταν εναντίον ε, περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Υπάρχει ένα πεδίο βολής, υπάρχει διαχείριση η οποία γίνεται μεταξύ της ε, αυτόνομης ε, κυβέρνησης ε, και υπάρχει και έλεγχος από την κυβέρνηση της Ισπανίας. Και έγινε και μία διαχείριση και έγιναν και έλεγχοι. Έχει περάσει όλους τους ελέγχους από το 1998 και μετά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. όταν χρησιμοποιείται το πεδίο βελής όλα τα κατάλοιπα συλλέγονται και ανακυκλώνονται για να είναι και σύνομα με όλους αυτούς τους ελέγχους αρμόδια για το πεδίο βολής είναι ε, η αυτόνομη περιοχή της ε, Βάρθενας και εκεί υπάρχουν 19 δήμοι, ε, ένα μοναστήρι, δύο κοιλάδες και είναι αυτή η αυτόνομη περιφέρεια που είναι αρμόδια και εκτός από μία περιοχή όλες οι υπόλοιπες από τις 21 περιοχές έχουν υπογράψει ε, την παράταση της ε, ε, λειτουργίας του πεδίου βολής. Αυτή είναι η αρμόδη και ποτέ δεν υπήρξε κάποια καταγγελία και διαμαρτυρία. Να σας πω επίσης ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε και στο Κογκρέσο και οι βουλευτές με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υποστήριξαν τη συνέχεια της δραστηριότητας του πεδίου βολής, 300, μία ψήφη υπέρ, 27 κατά και μία αποχή. Στην κυβέρνηση της Ναβάρα, η ομάδα που κυβερνά, που είναι η ομάδα της αριστεράς, με 26 ψήφους υπέρ, ζήτησαν να κλείσει το πεδίο βολής, αλλά δεν είναι αρμόδιοι για να κάνουν τέτοιο αίτημα. Και υπήρχαν 26 ψήφοι υπέρ και 24 κατά του κλεισίματος. Ε, οι ομάδες ε, που είναι πιο ε, ισχυρέ, Οι σοσιαλιστέ ε, και το Παρτίδο Ποπουλάρ, το Λαϊκό Κόμμα, ε, είναι υπέρ ε, τη παραμονή, του, αλλά δεν είμαστε εμεί οι αρμόδιοι. Οι αρμόδιοι είναι η περιοχή τη Μπάρθενα. και όλοι ζήτησαν να συνεχίσει, αλλά να υπάρχουν οι αυστηρότεροι περιβαλλοντικοί έλεγχοι για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω πολύ καλά γιατί βρέθηκε λοιπόν εδώ το θέμα, γιατί δεν υπάρχει καμία παραβίαση τη νομοθεσία. Επιπλέον οι αρμόδιε αρχέ επιθυμούν την παραμονή και εγώ λοιπόν θα ήθελα να ζητήσω Σα να κλείσει αναφορά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος ε, να λάβει το λόγο. Αυτό είχε μπει στην μέση διάταξη μετά από αίτημα της ΓΚΟΕ που δεν είναι καν παρούσα. Άρα δηλαδή θα πρέπει μάλλον να κάνουμε αυτό που είπε η Ρώσα και ως εκ τούτου να κλείσει αυτή η αναφορά. Από ό,τι βλέπω δεν διαφωνεί κανείς. Και πάμε στην επόμενη. Είναι η αναφορά 841 της Εβερίν Μπρέιτ ε, σχετικά με την κατάχρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών και την εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος μη γερμανών γονέων από το γερμανικό σύστημα οικογενειακού δικαίου από το Jugendamt. Έχουμε την Σεμπερίν Μπράιτ ε, μεταξύ μας και παρακαλώ να έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Αναφορών, αγαπητά μέλη της Επιτροπής. Να σας συστηθώ. Λέγομαι Σεβερίν Μπράιτ, είμαι Γαλλίδα υπήκος και έχω ένα αγοράκι που γεννήθηκε στη Γαλλία και είναι ηλικία 5 ετών. Έζησα στη Γερμανία, ζούσα στη Γερμανία όταν ο πρώην σύντροφό μου, Γερμανό υπήκο. Έλεγα λοιπόν ζούσαμε σε ένα κοινό σπίτι με τον σύντροφό μου και είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας και για να προστατευτώ και εγώ και το παιδί μου αποφάσισα να γυρίσω στη Γαλλία στους γονείς μου στα σύνορα ε, με κάθε νομιμότητα και με Γερμανίδα δικηγόρο γιατί σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο είχα την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού μου εκείνη τη στιγμή δεν ήμασταν παδεμένοι. και ε, το τονίζω αυτό είχα το γερμανικό νόμο στο πλευρό μου ο πρώην σύντροφός μου άρχισε ε, και ποινική διαδικασία και αστική στη Γερμανία και εκεί άρχισε ο μέγας εφιάλτης ο πρώην σύντροφό μου δεν είχε καμία επιμέλεια για το παιδί και δεν μπορούσε να ζητήσει να γυρίσει το παιδί πίσω μέσω της σύμβασης της Χάγης. Ε, και τον έβλεπε το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήματα και μου έστησε μία παγίδα και τον υποστήριξαν από το γερμανικό σύστημα, το οικογενειακό, το Jugendamt, που είναι ας πούμε το γερμανικό Υπουργείο ε, ε, Νεολαίας. το Jugendamt του έστειλε ένα πλαστό mail που του έλεγε ότι είχε την κοινή επιμέλεια μαζί μου, που ήταν τελείως και μου έρχεται ένα πρώτο γράμμα από γερμανικό δικαστήριο, επαναλαμβάνω και τονίζω, χωρί να έχει μεταφραστεί στη γλώσσα μου και μου λέει την άποψή μου. Πού θέλει το παιδί να μένει. Ε, σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο αυτό λέγεται Aufenthaltsbestimmungsrecht. Και είχα μια εβδομάδα για να απαντήσω ε, στη Γερμανία. Μια εβδομάδα σε ευρωπαϊκή χώρα σας φαίνεται λογική προθεσμία για τέτοια διαδικασία, για ε, διεθνή ε, ε, αίτηση για να μπορέσω εγώ να αμυνθώ σε κάτι που δεν είχα στη γλώσσα μου. Ε, ζήτησα μια συμβιβαστική συνάντηση μαζί με το παιδί και πήγα αφελώς γιατί δεν είχα τίποτα να φοβηθώ. Δεν μπορώ να σας πω τι έγινε ε, το 2017 8 Μαΐου. Ο δικαστής καταχράστηκε κάθε εξουσίας και κάθε δικαιώματος. Εγώ μπήκα με αποκλειστική επιμέλεια για το γιο μου εκεί, είχα νόμιμα μετακομίσει στη Γαλλία μαζί του και η δικαστής θα έπρεπε να θεωρήσει ότι είναι απαράδεκτο το αίτημα, τουλάχιστον να μην δώσει συνέχεια. Γιατί ε, ήταν αναρμόδιο το γερμανικό δικαστήριο, δεν έπραξε καθόλου κάτι τέτοιο. Τι έκανε, καταχράστηκε, ε, υπερεύει κάθε εξουσία χωρίς να συμφωνήσω και χωρίς να ζητήσει ο πατέρας εκ των υστέρων και μετά τη μετακόμισή μου έδωσε κοινή επιμέλεια. Αυτό το αίτημα δεν το είχε υποβάλει. Ε, το υπέβαλε στην ακροματική διαδικασία για να μου πάρει το παιδί και να το ε, πάει στη Γερμανία και έφυγα από το δικαστήριο τη μέρα των γενεθλίων του που έκλαινε τα πέντε χωρίς το παιδί μου, χωρίς τίποτα. Η Γερμανία απαγάγει, κλέβει παιδιά, γύρισα μόνη μου στη Γερμανία και το μόνο δικαίωμα που είχα ε, ήταν να του δώσω ένα φιλί και να του πω θα τα ξαναπούμε. Αυτά είναι ε, απάνθρωπα πράγματα για μια μητέρα. Η Γερμανία παραβιάζει κάθε ευρωπαϊκό κανόνα, ακόμα και τους ίδιους τους νόμους, για να παίρνει τα παιδιά των ανθρώπων. Ε, παραβιάζει την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μην φύγουν από τη Γερμανία τα παιδιά. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν μπορούν να ευτυχήσουν πουθενά αλλού τα παιδιά στην Ευρώπη, μόνο στη Γερμανία. Ε, ενώ το δικαστήριο ήξερε ότι είχα την αποκλειστική επιμέλεια όταν έφυγα, μου απήγαγαν το παιδί, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μου συνέβαινε κάτι τέτοιο το έτος 2017 σε χώρα ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με παγίδευσαν για να πάω στην ακροματική διαδικασία να χάσω το παιδί μου επιτόπου εγώ ζυγίζω τα λόγια μου, αλλά η Γερμανία, επαναλαμβάνω, μου έκλεψε και παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα και ενορχίστρωσε την απαγωγή του γιού μου. Και υφίσταμε τώρα και διπλή ποινή. Δεν φτάνει που ε, τρώω ξύλο τόσο καιρό, μου παίρνουν και το παιδί μου. Και μου αφαιρούν και όλα τα δικαιώματα. Βγήκα από το δικαστήριο χωρί να έχω το παραμικρό δικαίωμα στο παιδί. Δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα στην επίσκεψη. Θα πρέπει χωριστά να το ζητήσει δικαστικά. Πάρα πολύ γρήγορα λοιπόν κατάλαβα πώς δρούν τα γερμανικά δικαστήρια απέναντι σε γονείς που δεν είναι Γερμανοί. Το οικογενειακό σύστημα της Γερμανίας στοχεύει να κρατάει όλα τα παιδιά στη Γερμανία, παραβιάζοντας αν χρειαστεί και ε, ε, τον ευρωπαϊκό και το γερμανικό νόμο. Εμείς οι μη Γερμανοί γονείς ποτέ δεν πρόκειται να δικαιωθούμε στη Γερμανία, να βρούμε το δίκαιο μας σε δικαστήριο. Πώς γίνεται αυτό, πώς είναι δυνατό στην Ευρώπη. Νόμιζα ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία μας προστάτευε. Θέλω εδώ με την αναφορά αυτή να καταγγείλω ε, τη Γερμανία, την ασέβεια, τον τρόπο με τον οποίο παρακάμπτουν τους κανόνες, τους αγνοούν, ε, ε, ιδιαίτερα τον κανονισμό Βρυξέλλες 2Β, για να κλέβει τα παιδιά που έχουν διπλή ηθαγένεια ή είναι από γάμους. Είναι πολλοί οι γονείς που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα και το ξέρω υπάρχουν και ε, ενώσεις. Υπάρχει μια ένωση που ονομάζεται παιδιά όμοιροι. Ε, ε, μας καταστρέφουν τη ζωή. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και αναξιοπρεπή. Θα πρέπει να σταματήσει να αρπάζει τα παιδιά του κόσμου η Γερμανία και να μας τα γυρίσει πίσω. Πραγματικά σας εκλυπαρώ, βοηθήστε μας να σταματήσουμε αυτές τις δράσεις που είναι εγκληματικές ενέργειες. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας δραγίζει βέβαια και την καρδιά ε, και πολύ συγκινητικά όλα αυτά για όλους μας που βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή στην αίθουσα. Ε, καταλαβαίνουμε ότι είσαστε φορτισμένοι. Εμείς συμπάσχουμε με σας και με το γιο σας. Πολύ δύσκολη λοιπόν η κατάσταση. Βέβαια. Πρέπει τώρα να το δούμε το θέμα και να προσπαθήσουμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι ε, παρόλα αυτά με πολύ τρυφερά συναισθήματα, δύσκολη κατάσταση, κατάσταση και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην ε, Επιτροπή για να διαφωτίσει λιγάκι την κατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Προφανώς ε, και όλα αυτά είναι τραγωδίες, αλλά ξέρετε η Επιτροπή Αναφορών ε, δεν έχει πάρει ακόμα τις ε, δικές μας τις παρατηρήσεις. Θα έρθουν, θα τις πάρετε. Θα κάνω κάποια προκατακτικά σχόλια. Όπως είπε και αναφέρουσα, το δίκαιο ε, για ε, θέματα κοινής επιμέλειας ε, ασχολείται και με θέματα διασυνοριακά δεν ασχολείται μόνο με θέματα της απλής επιμέλειας και όπως σας είπα αρμόδιο δικαστήριο από αυτού θα ήθελα να πω ότι η Αποφάσισε του δικαστηρίου σχετικά με το που θα μείνει το παιδί, στην περίπτωση αυτή ε, εκδόθηκε μία εβδομάδα μετά την αναχώρηση της ε, μητέρας από τη Γερμανία. Αυτό δεν είναι κακή εφαρμογή του άρθρου 8, αλλά παραμένει μέσα στη διακριτική ευχαίρεια του δικαστηρίου να εξετάσει το δικαστήριο την περίπτωση. Και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ και σε μία παρεμφερή περίπτωση ε, περίπτωση Mercury 49 97-10 όπου το δικαστήριο αποφάσισε ότι εναπόκειται ε, στο Εθνικό Δικαστήριο να ορίσει τον τόπο διαμονής του παιδιού λαμβάνοντας υπόψη ε, όλα τα γεγονότα. Επίσης ε, θα ήθελα να πω ε, ότι στην περίπτωση αυτή ο πατέρας ε, δεν είχε την επιμέλεια ε, την στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη Γαλλία. Σε αυτή την άλλη περίπτωση. Και όσον αφορά τώρα τις απόψεις δικαστηρίου να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Οι Γερμανοί δικαστές πάντα θέλουν να ακούνε και την ίδια την άποψη των παιδιών σε θέματα που τα αφορούν, ακόμα και σε θέματα επιμέλειας και ακούγονται ακόμα και παιδιά των τριών ετών. Η Ευρωπαϊκή, Αρχή στηρίζει την... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την αρχή ότι το παιδί ε, θα πρέπει να εισακούει τα απόψή του αυτό βέβαια βρίσκεται και σε συμφωνία με την αναθεώρηση ε, του κανονισμού, ο οποίος περιλαμβάνει μία διάταξη όπου προβλέπονται υποχρεώσεις με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να εισακούεται η άποψη ενός ε, παιδιού που μπορεί βέβαια να εκφράσει τις απόψεις του. Σήμερα ήδη τα κρατημέλη ε, δεσμεύονται από τη Σύμβαση των ΗΠΑ για τα δικαιώματα του παιδιού που προβλέπει την υποχρέωση να εισακούεται εισακούεται η άποψη του παιδιού. Για να ολοκληρώσω ε, σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ότι υπάρχει παραβίαση ε, του ε, κοινοτικού δικαίου. Βεβαίω, σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα, γι' αυτό και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σε αυτή τη φάση, ακόμα και αν υπάρχουν ενδείξεις για παραβίαση του ε, ενωσιακού δικαίου. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συμβουλεύσουμε την αναφέρουσα ε, να εξαντλήσει όλα τα μέσα σε εθνικό επίπεδο. Η απόφαση, η του ε, γερμανικού δικαστηρίου είναι βέβαια προσωρινή μέχρι να υπάρξει η τελική απόφαση για την επιμέλεια και η αναφέρουσα θα πρέπει να αναφερθεί ε, σε θέματα κοινή ε, επιμέλειας αλλά να καταφύγει σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το περιεχόμενο της ε, απόφασης του Γερμανικού Δικαστήριου να σας πω ότι το οικογενειακό δίκαιο αναφέρεται το ότι και ορίζει ότι ο κανονισμός Βρυξέλλες 2 δεν ε, καθορίζει ότι όλα αυτά δεν εμπίπτουν στι αρμοδιότητε του ενωσιακού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την εφαρμογή μέσα από εθνικά δικαστήρια. Νομίζω ότι αυτό έχει αναφερθεί επανειλημμένα στην Επιτροπή των Αναφορών. Ω εκ τούτου το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πούμε ότι πρέπει κανεί να καταφύγει σε εθνικό δικαστήριο. Ε, ε, υπάρχουν και πληροφορίε για το πώς μπορεί κανείς ε, να αναζητήσει ε, αποκατάσταση και σε άλλα κράτη-μέλη. Θέλω να σας πω ότι εμείς δεν διαπιστώσαμε να υπάρχει παραβίαση του ενωσιακού δικαίου και γι' αυτό τη συμβουλεύουμε να αναζητήσει τη λύση σε εθνικό επίπεδο. Επειδή λοιπόν η αναφέρουσα θεωρεί ότι έχουν παραβιαστεί τα θεμελιώδη δικαιώματά της, ε, μπορεί και να καταφύγει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρόκειται να εργαστεί για την αναθεώρηση του κανισμού Βρυξέλλες 2. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Μαριάς, παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, το θέμα που έχει τεθεί έχει να κάνει με την διοικητική και δικαστική πρακτική που υπάρχει στο γερμανικό σύστημα, το οποίο έχει αποδειχθεί από συζητήσεις που έχουμε κάνει σε αυτήν εδώ την αίθουσα, ότι επιβάλλει διακρίσεις κατά των γονέων οι οποίοι δεν είναι Γερμανοί. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Θυμόσαστε εδώ, είχαμε φέρει γονείς οι οποίοι δεν ήταν Γερμανοί πολίτες και οι οποίοι είχαν καταγγείλει την πολιτική του Jugendamt, το οποίο χρησιμοποιούσε μια πρακτική διακρίσεων και ήταν πάντοτε υπέρ των γονέων που ήταν Γερμανοί πολίτες. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το δεύτερο είναι ότι όταν οι δύο γονείς ήταν αλλοδαποί, μη Γερμανοί, τότε το παιδί το έπαιρνε το Γιούγκενταμ. Επομένως εδώ η υπόθεση που έχουμε δεν έχει να κάνει τόσο με την εφαρμογή της οδηγίας για την δικαστική επίλυση διαφορών όταν έχουμε ένα μεικτό γάμο, αλλά εάν υπάρχει μια δικαστική πρακτική στα γερμανικά δικαστήρια, ούτως ώστε πάντοτε να εκδίδονται αποφάσεις υπέρ των Γερμανών πολιτών και εις βάρος των άλλων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι Γερμανοί. Και επομένως εδώ έχουμε παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης. Αυτό είναι το βασικό. Και η αρχή της δίκαιης δίκης περιέχεται στα θεμελιώδη δικαιώματα και στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως έχουμε μια νέα περίπτωση όπου όποια και να είναι τα ουσιώδη στοιχεία της υπόθεσης, το γεγονός ότι ο ένας γονέας είναι Γερμανός οδηγεί σε μια δικαστική απόφαση στα γερμανικά δικαστήρια υπέρ του γερμανού γονέα ανεξαρτήτως ουσιαστικά της ουσίας της υπόθεσης. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εγώ νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Και πρέπει να συγκεντρώσουμε και άλλες υποθέσεις. Και έχουμε όλο αυτό το υλικό. Και να ζητήσουμε πλέον από την Κομισιόν υπό αυτό το πρίσμα να δει αν γίνεται παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, αν τόσο το Jugendamt, η διοίκηση δηλαδή, όσο και τα δικαστήρια μεροληπτούν πάντοτε εις βάρος ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι Γερμανός. Αυτό είναι το θέμα. Και έτσι εκδίδουν αποφάσεις οι οποίες πάντοτε είναι υπέρ του γονέα ο οποίος είναι Γερμανός ανεξαρτήτως της ουσίας της ίδιας υπόθεσης. Εγώ νομίζω αυτό έχουμε μπροστά μας και επομένως σε αυτό το σημείο πρέπει να σταθούμε και γι' αυτό είχαμε συμφωνήσει να εκδικαστεί, να συζητήσουμε αυτή την αναφορά σύντομα διότι υπάρχει αυτή η διοικητική πρακτική και διότι έχει αφαιρεθεί το τέκνο ενός πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι Γερμανός. Αυτό πρέπει να εξετάσουμε και θα ήθελα και τη θέση των συναδέλφων από τη Γερμανία και του Πίτερ στο θέμα αυτό. Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές διότι εκεί πρέπει να σταθεί η Γερμανία. Δηλαδή να εξετάζει τόσο η διοίκηση, το Jugendamt, όσο και τα δικαστήρια αμερόληπτα κάθε υπόθεση και να μην μεροληπτεί υπέρ του γονέα που είναι Γερμανός. Αυτό είναι το θέμα και εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή υπόθεση και να συνεχίσουμε την έρευνα γύρω από το ζήτημα αυτό και να δούμε πώς μπορεί να αποφασίσουμε επί της ουσίας και να βοηθήσουμε τη λύση αυτής της υπόθεσης που έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν ζητήσαμε να εγγραφεί κατεπηγόντω αυτή η αναφορά στη σημερινή ημερήσια διάταξη, ακριβώ είχαμε επίγνωση αυτού του γεγονότο. ότι είναι κατεπηγούσα η κατάσταση και πραγματικά υποφέρει ε, ε, ε, αναφέρουσα και είναι και παράλογη η κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι ντρέπομαι από αυτά που ακούω. Δεν φταίει το δικό μας θεσμικό όργανο, αλλά όταν ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοια εικόνα δίνουν στους πολίτες για τόσο τραγικές περιπτώσεις τα θεσμικά όργανα. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα, πραγματικά. Και εμεί ως Επιτροπή Αναφορών θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας για να δοθεί άλλη απάντηση, άλλης ποιότητα και άλλης ε, φύση. Πέρα από τη συγκεκριμένη τραγωδία. <coughs> Ξέρουμε ότι δεν καθόλου καθόλου μεμονωμένη περίπτωση. Ε, τακτικά το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει. Και πέρα από την πραγματική συναισθηματική φόρτιση που το καταλαβαίνουμε, υπάρχει ένα διαρθρωτικό πρόβλημα εδώ. Ένας δημόσιος οργανισμός που φέρεται με τρόπο ε, που κάνει διακρίσεις εις βάρος των πολιτών. Αυτό είναι το θέμα. Όχι πως ερμηνεύουμε το τάδε άρθρο ε, των Βρυξελών ε, α ή β. Είναι εάν κάνει διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας δημόσιος οργανισμός. Και αν ισχύει αυτό πως δίνουν όλες οι αποχρώσεις ενδείξεις, δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρύβεται πίσω από την ερμηνεία ενός κανονισμού για να κάνει τα στραβά μάτια. Ε, υπάρχει το θέμα αυτό που αξίζει να εξετάσουμε και κατά πόσο γίνονται διακρίσεις. Είναι πάρα πολλές και δραματικές οι περιπτώσεις που ε, φτάνουν ε, στα χέρια μας και δεν μπορούμε να κοιτάμε από την άλλη μεριά όλα πάνε καλά. Και από πλευράς διαδικασίας επίσης, τι είναι αυτά τα πράγματα υπάρχει δίκαιο σύστημα όταν έχουμε γελίες προθεσμίες, αμετάφραστα νομικά κείμενα, αποφάσεις που λαμβάνονται στο φτερό ε, χωρίς ε, καμία προειδοποίηση στην ακροματική διαδικασία. Ακούμε ότι ε, τα αρμόδια δικαστήρια ακούνε και τα παιδιά. Και αν ο κίνδυνο είναι να πηγαίνει με το παιδί σου και να φεύγει χωρί αυτό, γιατί δεν έχει την επιμέλεια, τότε καταλαβαίνω ότι θα τεθεί διαφορετικά το θέμα να ε, μιλούν στα δικαστήρια και τα παιδιά. Λοιπόν, η δίκη, η δίκη για μένα είναι άλλο πράγμα. Χρειάζεται πολύ μεγάλη εξέταση πέρα από την απλή ερμηνεία ενός κανονισμού Βρυξέλλες 2. Πώς λειτουργεί το Jugendamt, να το κοιτάξουμε αυτό ε, βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων και των διακρίσεων και το σεβασμό της οικογενειακής βίας. Αυτό, ε, του οικογενικού βίου, συγγνώμη. Έχουμε αρμοδιότητες, έχουμε ιδρυτικά κείμενα και από τον ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τώρα αμφισβητούνται. Και θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί το Γιουγέντα. Παρακαλώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει περισσότερα και να το ψάξει περισσότερο. Εμείς ως Επιτροπή Αναφορών να ασχοληθούμε ξανά με το θέμα αυτό και να το μάθει και η γερμανική κυβέρνηση. Ναι, ευχαριστώ. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την αναφέρουσα γιατί μας παρουσίασε για πολλωστή φορά μια υπόθεση που αφορά το Jugendamt και θα ήθελα να επισημάνω και το γεγονός ότι πάνω από 10 χρόνια φτάνουν εδώ στην Επιτροπή Αναφορών αναφορές ε, που ε, αφορούν σοβαρές καταγγελίες όσον αφορά τη συμπεριφορά του Jugendamt. Ε, διακρίσεις ε, ενώπιον ε, πολιτών και γονέων που δεν είναι γερμανικής υπηκότητας. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την πρώτη αναφορά, αλλά γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά ότι το μέσο αυτό δεν είναι απεικόνηση του πραγματικού προβλήματος, είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. αν σκεφτεί κανείς ε, τον αριθμό των πιθανών περιπτώσεων. Εδώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι όσον αφορά τον ε, ε, κανονισμό Βρυξέλλες 2, διότι θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εφαρμογή του νέου κανονισμού και η τροποποίησή του κινδυνεύει να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τα πράγματα για μη Γερμανούς πολίτες. Διότι καταργείται το Ινστιτούτο το οποίο αποτελεί πηγή έμπνευσης του γεγονότος ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ ε, αρχών, δικαστικών και διοικητικών αρχών και αυτό θα ήταν θετικό, αλλά ελοχεύει ο κίνδυνος να γίνονται αυτομάτως οι διακρίσεις ακριβώς λόγω της εφαρμογής μέτρων ε, ε, μέσω της παρέμβασης του Jugendamt. Και αυτό βασίζονται σε μια πολύ διόρυθμη ε, ερμηνεία του ε, να γίνει ότι είναι ε, καλύτερο για το παιδί, για τον ανήλικο. Και η απάντηση του Ομοσπονδιακού Υπουργού ε, στην οικογένεια ε, αρμοδίου για θέματα οικογενεία σε όσα αιτήματα έχουμε κάνει στο παρελθόν για την προστασία των ανηλίκων. Η έννοια τη προστασία του ανηλίκου στη γερμανική νομοθεσία είναι πάρα πολύ αμφίσιμη. Δεν ορίζεται βάση τη νομοθεσία, ε, αλλά ε, βάση τη νομολογία. Και αυτό ε, σημαίνει ότι υπάρχει, ναι, μεν αυτό το υποτιθέμενο συμφέρον του παιδιού και θα μπορούσε να ισχύει εδώ ακόμα και το πιο παράδοξο για την προστασία και το συμφέρον του παιδιού. ενώ κανονικά θα έπρεπε να μην υπάρχει διάκριση από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη. Ε, αν γίνει λοιπόν αυτή η τροποποίηση, ο κίνδυνο ε, να επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά και βάσει των τελικών συστάσεων ε, της ομάδας εργασίας για την ευημερία των ανηλίκων και νομίζω ότι θα μπορούσαμε ίσως να στείλουμε άλλη μία επιστολή στον Ομοσπονδιακό Υπουργό Αρμόδιο για θέματα οικογένειας στη Γερμανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρτών. Ευχαριστώ. Δεν ναι, υπάρχει κανείς καλύτερος από εσά, ε, κυρία Πρόεδρε, που γνωρίζετε τις εργασίες της Επιτροπής, που ξέρετε, όπως και οι υπόλοιποι, ότι έχουμε ασχοληθεί με δεκάδες τέτοιες υποθέσεις του Γιούγκενταμ και δεν ξέρω καμία περίπτωση, ούτε μία, στην οποία ε, να μην γίνεται διάκριση κατά του μη Γερμανού ε, γονιού και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι μη Γερμανοί ε, γονεί είναι αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν τον νόμο, κανένα δεν σέβεται τον νόμο και οι μόνο Γερμανοί είναι ονοματάκε πολίτε. Ε, επιτρέψτε μου να έχω κάποιε αμφιβολίε από αυτού. Ε, ακόμα και εδώ στην αίθουσα νομίζω πριν από ένα χρόνο ε, και εσείς είχατε επιμείνει πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε για να έχουμε τη δυνατότητα να ε, μιλήσουμε με το Γιούγκενταμ. Ήρθαν Είπαν αυτά που γνωρίζουμε όλοι, ότι είμαστε εμεί εδώ για να προστατεύσουμε το συμφέρον του παιδιού. Το θυμάστε, εκεί πίσω καθόντουσαν. Ήταν ένα παιδάκι, ή μάλλον ε, ένα νέο 18 ετών Πολωνό, που είχε βιώσει αυτή την κατάσταση ε, και του δώσατε το λόγο, θα το θυμάστε, και ο νέος αυτό άνθρωπος είπε στο Γιούγκεντα αυτό είναι ψέμα αυτό. Εγώ ε, είμαι μεταξύ αυτών των νέων παιδιών που θέλω να βλέπω την Πολωνή μητέρα μου και εσείς μου το απαγορέψατε. Υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο αφορά και την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων. Αυτό αντίκειται στην νομοθεσία και το ε, πνεύμα τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και αυτό είναι και το λάθο τη κυρία Μπράθ, Bright. Ε, ε, λάθος, όχι σφάλμα. Ε, μίλησε με ιδιαίτερο πάθος, διότι όταν ένας γονιός χάνει το παιδί του, πώς αλλιώς να τα πει. Το λάθος της είναι ότι εμπιστεύτηκε τη δικαιοσύνη και τα δικαστήρια και την παγίδευσαν. αν είχε μείνει ήρεμα στη Γαλλία θα ήταν με το παιδί της σήμερα τι να κάνουμε εμείς οι Ευρωπαίοι βουλευτές που δεν είμαστε Γερμανοί. Τι να ζητάμε από τους μη Γερμανούς γονείς να πηγαίνετε στη Γερμανία να κλέβετε τα παιδιά σας και να κάνετε αυτό που κάνουν. Αυτό θέλετε. Θέλετε να κάνουμε αυτό το πράγμα διότι δεν γνωρίζω ούτε μία περίπτωση ε, να μου βρείτε από την Κομισιόν μία περίπτωση στην οποία να δόθηκε δίκιο στο μη Γερμανό γονιό. Και εγώ που είμαι από την περιοχή της κυρίας ε, Μπράιτ γνωρίζω δεκάδες τέτοιε υποθέσεις. Ε, δεν υπάρχει τήρηση τη νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση και η Γερμανία το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει ήδη καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι πρέπει να καταγγείλουμε την υποκρισία των κρατών μελών. Ε, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κρυφή δύναμη, αυτή η κρυφή εξουσία στη Γερμανία, γιατί ακόμα και η δική μου κυβέρνηση, στην οποία αποτάθηκαν και ζήτησαν να διαχειριστούμε την κατάσταση και μίλησα για την υπόθεση τη κυρία Μπράι. Και ξαφνικά όταν μιλάμε για το Jugendamt, ξαφνικά είναι λεπτό ζήτημα και δεν μπορούμε να το συζητάμε. Καταγγέλω λοιπόν εδώ την υποκρισία των κρατών μελών και θα ήθελα να ξέρω ποιε είναι αυτέ οι σκοτεινέ δυνάμει και τι εξουσία έχουν. Πού βρίσκεται αυτή η εξουσία πραγματικά γιατί εγώ δεν ε, τη βλέπω. Παθιάζεστε με αυτά τα θέματα και εγώ παθιάζομαι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε λίγο να είμαστε ήρεμοι, διότι δεν ε, ε, βοηθά και κανέναν να επενδύουμε τόσο πολύ τα συναισθήματά μας στο θέμα αυτό. Είναι μία αναφορά σαν όλες τις άλλες. Ο Πέτερ. Από μου τώρα το λυπηρό ποιο είναι, το είπαν και οι συνάδελφοι. Πριν από 10 χρόνια ε, είχαμε κάνει ακρόαση, είχε έρθει εκπρόσωπο στο Jugendamt, έχουμε κάνει ομάδα εργασία στην Επιτροπή Αναφορών. Ποιο είναι το πρόβλημα σε τέτοιε περιπτώσει, καταρχήν. Ότι δεν είναι ε, κεραυνός ενεθρία ε, και δεν είναι σε φιλικό περιβάλλον. Ε, ε, είναι άνθρωποι που αγαπιούνται, μετά χωρίζουν, μετά έχουν εντάσεις μεταξύ τους και συγκρούονται και σε αυτή την περίπτωση. Εδώ συμμετέχουν συνήθως τρεις ενδιαφερόμενοι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο άντρας, η γυναίκα και το παιδί. Τώρα ακούμε τη μία πλευρά και δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Σε καμία περίπτωση. Και όσο δύσκολα και να είναι αυτά και όσο παραξικάρδια και να είναι, θα πρέπει να είμαστε και ειλικρινεί και τίμοι στην Επιτροπή μα και να λέμε πού μπορούμε να βοηθήσουμε και δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Εδώ είναι θέματα βαθιά περίπλοκα νομικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει, η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορεί να βοηθήσει. Και δεν το θεωρώ και δίκαιο απέναντι στου αναφέροντε να αφήνουμε ανοιχτή μια αναφορά. Τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επί τη ουσία δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον αναφέροντα. Η κορφή του παγόβουνου, λέτε, είναι το Γιούγκενταμ. Στο 99% των περιπτώσεων το Jugendamt ασχολείται με ενδογερμανικά θέματα. Είναι σαφές και αυτό εντός της Γερμανίας. Και το 1% αφορά, ε, όπως φαίνεται, ε, αφορά ε, μη ε, Γερμανούς πολίτες, ε, Πολωνούς, Γάλλους, ε, υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης. Δεν θέλω να τα επαναλάβω όλα αυτά. Τα έχουμε συζητήσει, ε, επανειλημμένα, εξαντλήσει. Το βασικό πρόβλημα για μένα ε, σε περίπτωση σύγκρουσης είναι πρώτον η ίση Γιατί έχει περισσότερα δικαιώματα ο πατέρα ή η μητέρα όταν τσακώνονται οι δύο. Και, τα δύο, και στη διένεξη αυτή οι νομικοί έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και υπάρχει και η σύμβαση της Χάγης σε περίπτωση ε, σύγκρουσης θα πρέπει να είναι προς το συμφέρον του παιδιού και να παραμένει εκεί που είναι το κέντρο της ζωής του να διαμένει το παιδί. Και σε πολλές περιπτώσεις είναι η χώρα που έχει μεγαλώσει. Αυτό μπορεί να μην το καταλαβαίνουν εύκολα οι ενδιαφερόμενοι, αλλά εμείς είμαστε Επιτροπή Αναφορών, δεν είμαστε δικαστήριο. Επιλεκτικά ακούμε τον αναφέροντα αναγκαστικά δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα, δεν είμαστε δικαστήριο, δεν έχουμε νομοθετικές αρμοδιότητες ίδια του νόμου. Το παραλαμβάνω, αλλά είναι ειλικρίνεια να λέμε στον αναφέροντα πού μπορούμε να βοηθήσουμε. Εδώ μπορούμε να σε βοηθήσουμε, εδώ δεν μπορούμε. Και στι περισσότερε περιπτώσει είναι τόσο περίπλοκα νομικά ζητήματα που πραγματικά χρειάζεται να το διεκδικήσει αυτό κανεί δια τη νομική οδού και όχι δια τη Επιτροπή Αναφορών. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στανόκα. Yes, thank you. Also, I came later. Ευχαριστώ. Ε, καθυστέρησα κι εγώ να μπω από την Επιτροπή Επασχόλησης έρχομαι και θα ήθελα να σας δώσω μερικές ε, από τις σκέψεις μου γιατί είμαι μέλος στην ομάδα εργασίας ε, για την ευημερία των ε, παιδιών. έχω και εμπειρία από προηγούμενες αναφορές και υποθέσεις για το Γιούγκεντα. Μακρά εμπειρία έχω. Τα τελευταία εννέα έτσι εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Κύριε Γιάρ, δεν συμφωνώ με αυτά που λέτε το τελευταία, ότι οι διασυνοριακές περιπτώσεις δεν είναι τόσο απλές δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη λύση του συμφέρον του παιδιού να παραμένει στη χώρα που μεγάλωσε που γεννήθηκε δεν είναι τόσο απλό αυτό ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Το παιδί δεν ανήκει σε κράτη. Όταν μιλούμε για πολιτικές θέσεις θα πρέπει να έχουμε όλα αυτά υπόψη μας. Κοίταξα τις συστάσεις εγώ. Και πώς να σας το πω. Φοβάμαι. Η σύσταση να στείλουμε μια επιστολή τι επιστολές να στείλουμε και σε ποιον. Στις γερμανικές αρχές, στις γαλλικές αρχές γιατί να στείλουμε επιστολή. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε ε, εσείς που το προτείνετε γιατί να στείλουμε επιστολή στις γαλλικές αρχές. Εγώ θα πρότεινα απλώς για να μην επαναβάλλω τα επιχειρήματα να μην ανοιχτεί η αναφορά αυτή και να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή περισσότερη πληροφόρηση. Τη επιστολή να τη στείλουμε στη γερμανική ε, κυβέρνηση, ιδιαίτερα στο Jugendamt. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, δεν έχω άλλους ομιλητές στον κατάλογό μου και θα ήθελα τώρα να σας δώσω το λόγο στην αναφέρουσα για δύο λεπτά, δύο επιπρόσθετα λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς για να διευκρινίσω στους Γερμανούς, ο πρώην σύντροφό μου μου έστελνε μηνύματα στα οποία μου έλεγε ο ίδιος ότι θα πρέπει να επιστρέψω στη Γαλλία. Αυτό έκανα γιατί αυτό μου το ζήτησε είχα ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Γαλλία. Για μένα λοιπόν το γερμανικό δικαστήριο ήταν αναρμόδιο. Παραβίασε τα θεμελιώδη δικαιώματα, το άρθρο 8 του ε, Βρυξέλλες 2. Το παιδί πήγαινε σχολείο στη Γαλλία σε ε, ε, προσχολική αγωγή και επομένως είχα ξεκινήσει μια νέα ζωή στη Γαλλία και επομένως αρμόδιο έπρεπε να είναι το γαλλικό δικαστήριο. Παραβίασαν το δίκαιο και παραβίασαν το δίκαιο σε αυτό το επίπεδο διότι θεώρησαν ότι είναι δική του αρμοδιόθεση ε, αρμοδιότητα παραβίασαν το δίκαιο διότι άλλαξε έρευνα στην διάρκεια της ακρόασης. Ο, πατέρας είχε ζητήσει την κυδαιμονία γιατί δεν είχε την επιμέλεια στη διάρκεια της ε, ακρόασης ε, και αυτό είναι παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου και έκανε νέο αίτημα στη διάρκεια της ακρόασης. Δεν μπορεί να καταθέσει νέο αίτημα στη διάρκεια ακρόασης. Το κείμενο δεν ήταν μεταφρασμένο και υπήρχε και ένα μνημόνιο το οποίο κατατέθηκε την ημέρα της ακρόασης. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ένα υπόμνημα σε αυτή την περίπτωση. Ε, δεν μπορούσα εγώ να έχω και υπόμνημα να απαντήσω. Ε, λοιπόν, πέρα του γεγονότο ότι παραβίασε το ευρωπαϊκό δίκαιο, παραβίασαν και τη δική του νομοθεσία η Γερμανία. Αυτά ευχαριστώ. Και πραγματικά, αν κλείσει η αναφορά μου, η Γερμανία θα μπορεί να συνεχίσει να κλέβει και άλλα ε, παιδιά σαν το δικό μου, γιατί έχουν πάει πολύ παραπέρα από ό,τι συνήθω. Εγώ δεν ήμουν απαντρεμένη, είχα αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού και σημαίνει ότι αν κλείσετε την αναφορά μου από εδώ και σε, πέρα θα συνεχίσουν να κλέβουν παιδιά από μη γερμανού γονιού και οποιοδήποτε μη γερμανό θα συνεχίσει να προσφεύγει στη Γερμανία, αλλά ποτέ δεν θα ξαναπάρουμε τα παιδιά μα πίσω. Ποτέ. Σα ευχαριστώ πολύ. Και κάτι ακόμα να το διευκρινίσω, γιατί εγώ ζήσω, σε περιοχή των συνόρων και μου λένε ότι ήμουν στη Γερμανία, θέλω να διευκρινίσω ότι στα γερμανογαλλικά σύνορα υπάρχουν πολλοί Γερμανοί που ζουν από τη γαλλική πλευρά και αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί όταν ζουν στη Γαλλία πάνε στο παιδί, παίρνουν το παιδί του και πάνε από την άλλη πλευρά του συνόλου στη Γερμανία, τότε το Γιούγκεντα λέει ότι είναι πολύ αργά, τα παιδιά βρίσκονται σε γερμανική επικράτεια, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, το παιδί ε, είναι αρμοδιότητα του γερμανικού δικαστηρίου. Επομένω, είτε βρισκόμαστε στη Γαλλία είτε βρισκόμαστε στη Γερμανία, το παιδί επιστρέφει στη Γερμανία και επιστρέφει στη γερμανική επικράτεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Εγώ σας ευχαριστώ. I think we need to conclude this. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσει εδώ αυτό το θέμα. Άκουσα τους συναδέλφους να λένε ότι θέλουν να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Κανείς δεν θέλει να κλείσει. Ωραία. Θα την κρατήσουμε ανοιχτή. Και η πρότασή μου είναι να στείλουμε την αναφορά ε, στο, στο Intergroup, τη διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των ανηλίκων, για να το κοιτάξουν και από άλλες σκοπιές το ίδιο θέμα. Έχετε τίποτα άλλο προτείνετε. Μιλήσατε όλοι πολύ, αλλά δεν προτείνατε και κάτι συγκεκριμένο. Ο κύριος Μαριάς. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Συμφωνώ να πάει στο γκρουπ ε, που ασχολείται με τα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού. Προτείνω. Πρώτα απ' όλα πρέπει να στείλουμε μία επιστολή στο Jugendamt διαμαρτυρίας για την διοικητική πρακτική που έχει, ούτω ώστε πάντοτε μεροληπτεί υπέρ των Γερμανών πολιτών. Και επιπλέον να ζητήσουμε από την Κομισιόν στοιχεία, δηλαδή στις, να μας φέρει στοιχεία αν στις δίκες στα δικαστήρια όπου υπάρχουν υποθέσεις μεταξύ Γερμανών πολιτών και μη Γερμανών πολιτών πόσες φορές έχουν κερδίσει τις υποθέσεις αυτοί που δεν είναι Γερμανοί πολίτες και ποια είναι η διοικητική πρακτική του Γιούγκενταμ. Και με βάση αυτά τα στοιχεία να ετοιμάσει η Κομισιόν ένα φάκελο για την περίπτωση παραπομπής της Γερμανίας στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διακριτική μεταχείριση έναντι των υπολείπων πολιτών ως διοικητική πρακτική. Αλλά αυτό να γίνει από την ίδια την Κομισιόν η οποία να μαζεύσει τα στοιχεία και να επαναφέρουμε αυτή την υπόθεση κάποια στιγμή για να μας ενημερώσει που βρίσκεται. Αν το αφήσουμε μόνο στις προτάσεις που λέτε δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το Γιωγενταμ και τα δικαστήρια στη Γερμανία θα συνεχίσουν να μεροληπτούν. Έχουμε υποθέσεις πάρα πολλές και Ελλήνων πολιτών και άλλων πολιτών που έχουν υποφέρει από την λειτουργία του Γιούγκενταμ. Η Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα κάνει αρκετές προτάσεις, ε, πέραν του γεγονότος ότι ζητώ να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή, εγώ πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να γίνει, ε, γιατί όχι να πάει και στην διακομματική ομάδα, στο Intergroup, συμφωνώ απολύτω με την πρόταση του συναδέλφου Μαριάς, Μαριά, να ζητήσουμε πέραν των αναλύσεων που μας έγιναν ε, σήμερα, ε, διότι είναι ανεπαρκής, να μα κάνουν μια δεξιοδική ανάλυση. Έχουμε πάρα πολλές υποθέσει με θέμα το Jugendamt. Ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση βέβαια και τις πληροφορίες που διαθέτουν, τώρα είναι θεμελιωμένες ή όχι αυτές οι ε, δηλώσεις, αυτοί οι ισχυρισμοί, ε, φαίνεται ότι υπάρχει διάκριση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό, επομένως θα πρέπει να το διερευνήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δει τι έχει με βάση τα πτά στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και να δει αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση ε, ή όχι. Και αν όντω διαπιστωθεί διακριτική μεταχείριση δεν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση, να δούμε τι κάνει το Jugendamt και αν όντω γίνεται διακριτική μεταχείριση. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και το εξή μπορούμε να δούμε και το θέμα της δίκαιης δίκης εδώ, όταν βλέπουμε ότι δεν υπήρχε μετάφραση, πολύ σύντομες προθεσμίες, ο τρόπος με τον οποίο έγινε αυτή η δίκη. Ε, για μένα λοιπόν, ε, ε εάν επαληθευτεί, θα το εξετάσουμε, ε, μήπως ε, έχουμε το δικαίωμα να δούμε και τι γίνεται και το ε, θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και μήπως παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα σε αυτή την περίπτωση. Θέλω λοιπόν να υποβάλουμε το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης θα ήθελα πέραν αυτού εμεί ω Επιτροπή να ε, ε, στείλουμε αίτημα στην ε, νέα γερμανική κυβέρνηση για το θέμα του Γιούγκενταμ. Αυτά λοιπόν προτείνω για τη συνέχεια τη συγκεκριμένη αναφορά. Η Ελεονόρα. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω ότι στην παρέμβασή μου Ανέφερα και την επιστολή στο Γερμανό Ομοσπονδιακό Υπουργό. Αυτό προτείνω και εγώ και υποστηρίζω λοιπόν ακράδαντα την πρόταση των Σοσιαλιστών Δημοκρατών και του ECR. Εκτός μικροφώνου κυρία Ζδάνοκα. Ωραία, λοιπόν, θα κάνουμε το εξή. Ακούσαμε πολύ προσεκτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δήλωσε σαφέστατα ότι δεν υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, λοιπόν, να πάμε πάλι στην Επιτροπή και να τη ρωτήσουμε κατά πόσο υπάρχει παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, όταν μα είπαν σαφέστατα ότι δεν υπάρχει παραβίαση ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση είναι να παραμείνει αναφορά ανοιχτή, να στείλουμε επιστολή στο Jugendamt για τη διαδικασία, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος ε, Μαριάς για τη διοικητική διαδικασία. Αυτό σίγουρα μπορεί να γίνει. Και από εκεί και πέρα να στείλουμε και επιστολή στις γαλλικές αρχές και να ζητήσουμε να υποστηρίξουν όσο μπορούν ε, ένα Γάλλο υπήκο, ο οποίος ε, είναι θύμα σε αυτή την περίπτωση και να στείλουμε και επιστολή τις γερμανικές αρχές να πούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουν τη λειτουργία του Jugendamt. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Επιπλέον, Τατιάνα, τι άλλο θες. Σε συνέχεια της πρότασης της κυρίας Ροζιέρ, να μας δώσουν και πληροφορίες. Και ο κύριος Μαριάς πρότεινε κάτι αντίστοιχο για την ανάλυση των διασυνοριακών υποθέσεων Από ποιον ζητάμε πληροφορίες. Πρέπει να υπάρχει κάποια μελέτη. Ε, τώρα βέβαια δεν μπορούμε να ε, παραγγείλουμε μελέτη. Φαντάζομαι όμως οι γερμανικές αρχές, ο Υπουργός έχει στατιστικά στοιχεία για αποφάσεις ε, δικαστηρίων για γονική μέρημνα και επιμέλεια σε διασυνοριακές υποθέσεις αυτό που είπε ο κύριος Μαρτάν, ότι το 100% είναι υπέρ των Γερμανών. Ε, αυτή την αίσθηση έχει, αλλά χρειαζόμαστε και στατιστικά στοιχεία. ποτέ δεν πρόκειται να αποκαλύψουν τέτοια στατιστικά στοιχεία. Μπορεί να στείλουμε επιστολή, όπως είπε η κυρία Ροζιέρ, και να πούμε ότι θέλουμε να μελετήσουν τη λειτουργία του Jugendamt σε σχέση με αυτό η Βερζινή. Ε, Καλά, έχουμε κάποιες περιπτώσεις που μας αφήνουν να καταλάβουμε ότι υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Είναι φυσιολογικό ε, να θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει αρμοδιότητες για να εξετάσει τι γίνεται αν είναι αυτή η πραγματικότητα, αν δεν είναι πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις διακριτικών πρακτικών. Ε, όχι διάβασα εντάξει τι λέει το γράμμα του κανονισμού Βρυξέλλες 2 και είμαστε εντάξει. Έχουμε ολόκληρη στίβα φακέλων. Εκ πρώτη όψεω, εμείς βλέπουμε ότι μεροληπτούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τόσα μέσα και τόσου πόρου αν το εξτάσει ε, θα το διαπιστώσει όλη αυτή τη μάζα αν ε, κάνουν διακρίσεις, φυσιολογικό είναι να το ζητάμε. Ε, το ζήτησε νομίζω και ο κύριος Μαριάς προς την κατεύθυνση αυτή, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάση των διασυνοριακών, ε, δεν είναι γερμανική δικαιοδοσία στη γερμανική επικράτεια, είναι διασυνοριακές υποθέσεις, να διαπιστώσουμε αν υπάρχει όχι διακριτική στάση υπέρ των Γερμανών και κατά των μη Γερμανών γονέων αν μη τι άλλο, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Να δούμε πόσε είναι οι περιπτώσει. Επανειλημμένα έχουμε προβληματικέ ε, υποθέσει εδώ. The Commission wants to come in here. Please go ahead. Η Κομισιόν θέλει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία ότι ο Βρυξέλλες 2α δεν ε, περιλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για συλλογή στατιστικών δεδομένων σε διασυνοριακές υποθέσεις, αλλά η αναθεώρηση ε, περιλαμβάνει πρόταση στο άρθρο 79, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να συλλέγουν τα κράτη-μέλη πληροφορίες ε, για τον αριθμό των αποφάσεων, και την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες, Βρυξέλλες 2α. Και αυτό φυσικά θα βοηθήσει να έχουμε στοιχεία για το θέμα και να μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία και ορισμένες φορές είναι πολύ δύσκολο, διότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο δικαστηρίου. Εάν από εκεί και πέρα δεν συλλέγονται στοιχεία όσον αφορά το ε, κατά πόσον το συμβαλόμενο μέρος είναι από διαφορετική χώρα, ε, τα στοιχεία μπορεί και να μην υπάρχουν καν. Ευχαριστώ. Η Έλα. Δεν χρειάζεται νομική βάση στη Βεξέλλες 2α για να κάνει έρευνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει υποψία ε, ότι τα κράτη-μέλη δεν ε, τηρούν τις συνθήκες. Είναι θεματοφύλακες των συνθήκων και αν λείπει στατιστική βάση, νομίζω ότι ο αριθμός των υποθέσεων που μας έχουν απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή Αναφερών ούτως ή άλλως θα έχουν αρκετά μεγάλο φάκελο. Θα πρέπει λοιπόν να ερευνήσουμε τι γίνεται σε περίπτωση ε, ε απουσία στοιχείων και δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε τον Βεξέλλες 2α γι' αυτό. Η Ελεονάρα Εύη. Θα ήθελα να κάνω μια άλλη πρόταση. Πιστεύω ότι επειδή είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, ίσως θα έπρεπε το θέμα να συζητηθεί και στην Ολομέλεια με προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να υπάρχει και ψήφισμα. Πιστεύω ότι έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορεί να ανάψει πλέον αυτό το πράσινο φως και παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για να συνεχίσει, να πιέσουμε εμείς τα πράγματα γιατί από πολιτικής πλευράς θα πρέπει να λάβουμε θέση σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Να υπενθυμίσω ότι βάσει των κανόνων αυτής της Επιτροπής ε, δεν αλαμβάνουμε εμεί αποφάσεις ε, για ε, θέματα στην Ολομέλεια και προφορικές ερωτήσεις. Αυτή είναι η συζήτηση των συντονιστών. Έχετε τη δυνατότητα να το θέσετε στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, μπορείτε να το συζητήσετε με τους αδέλφους, αλλά όχι στην τακτική συνεδρίαση. Ο κύριος Μαριάς. Στην αναφορά που έχουμε. Άρα λοιπόν Όλες οι προτάσεις έχουν κατατεθεί. Απλά συμπληρώνω αυτό που είπαμε από την αρχή. Η, ζητούμε ξανά εμείς από την Κομισιόν να, να δει εάν υπάρχει διάκριση με βάση τον κλασικό όρο της συνθήκης, η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ηθαγένειας. Αυτή είναι η λειτουργία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένου το Jugendamt ως διοικητική πρακτική Έχουμε όλα τα στοιχεία που δείχνει ότι παραβιάζει τη βασική αρχή λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηθαγένειας. Αυτό λοιπόν να το εξετάσει, να δει αν υπάρχει αυτή η διοικητική πρακτική, να έρθει να ενημερώσει την Επιτροπή μας και από την ώρα που υπάρχει αυτή η διοικητική πρακτική πρέπει μετά να προχωρήσει σε αυτό που λέει η συνθήκη. Να παραπέμψει στη Γερμανία για παραβίαση της συνθήκης λόγω διακρίσεων. Αυτό είναι. Αλλά εμείς ζητούμε από την Κομισιόν να το ελέγξει αυτό. Υπάρχουν τα στοιχεία σε αυτή τη βάση και όχι με βάση ε, το Βρυξέλλες 2. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Και έχουμε πάρα πολλά στοιχεία. Ξέρουμε τι κάνει το Γιούγκενταμ. Ας μας φέρει μια περίπτωση όπου ένας πολίτης που δεν είναι Γερμανός έχει κερδίσει μια υπόθεση ή στο Γιούγκενταμ ή στα δικαστήρια. Αυτή είναι η ουσία. Okay. Κοιτάξτε, ωραία. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ αυτό το θέμα. Έχουμε αφιερώσει τόσο χρόνο. Θα προχωρήσουμε ω εξή. Να κρατήσουμε ανοιχτή την ε, αναφορά. Θα στείλουμε επιστολή και στο Jugendamt και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το κοιτάξει. δεν είναι σύνηθες αυτό το αίτημα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι κάτι που υπερβαίνει αυτό το πλαίσιο και θα πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς. Ε, βάσει του συγκεκριμένου περιστατικού ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το εξετάσει. Πρέπει να ξαναπώ ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Εδώ είναι συνεδρίαση επιτροπών. Και εδώ μιλούμε, πετάμε ονόματα, μιλάμε για παιδιά, για ανθρώπους που δεν είναι παρόντες. Εντάξει, μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για την τροποποίηση του κανονισμού 883 και 987 του 2009 και λοιπά. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σολεδάθ Καμπεθόν Ρουίθ. Καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας και πάλι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ε, Δεκέμβριο του 2016 έκανε πρόταση κανονισμού για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης ε, με στόχο την απλούστευση και την αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας που βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενισχύσουμε την αρχή της ευρωπαϊκής ε, ηθαγένειας του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, άρα χρειάζεται να δούμε και τα κοινωνικά δικαιώματα. Στη γνωμοδότησή μας εμείς επικεντρωθήκαμε σε τέσσερα σημεία αναπηρία, υγεία, ε, ανεργία και συντάξεις, αλλά κυρίως τα δύο πρώτα. Για τις συντάξεις θεωρούμε γενικά ότι ο κανονισμός είναι καλός και έχει δίνει καλή λύση, αλλά για την ανεργία ε, ζητήσαμε να ε, εξομοιωθεί με το σύστημα των συντάξεων σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των δικαιωμάτων. Και επίσης ζητήσαμε από τρίμηνο να γίνει ένας μήνας το δικαίωμα ε, σε επίδομα ασφαλείας, ε, σε επίδομα ανεργίας, συγγνώμη. Όταν φεύγει κάποιος από τη χώρα του, όχι μετά από ένα τρίμηνο, αλλά μετά από ένα μήνα να έχει δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας. Και επίσης αυτό περιορίζεται με βάση το δικαίωμα που έχεις θεμελιώσει και σου έχουν αναγνωρίσει στη χώρα σου. Αλλά δεν θα πρέπει να περιορίζεται αυτό λοιπόν όταν πηγαίνεις σε άλλη χώρα ως προς το χρόνο ε, που είσαι δικαιούχος ε, του επιδόματος ανεργίας ε, όταν έχεις το δικαίωμα αυτό στη χώρα σου. Για την αναπηρία, τι ζητήσαμε γίνεται λόγο στον κανονισμό στον Ευρωπαϊκό Χάρτη για την αναπηρία, αλλά εμείς επιπλέον ε, συγγνώμη, στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρία, ε, αλλά ζητούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστεί η Σύμβαση ε, των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. δεν έχουμε λοιπόν δικό μας ορισμό, ακόμα δεν υπάρχει συνένεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ορισμό αυτό. Γιατί το ζητούμε εμείς, διότι για να είναι τα δικαιώματα ακριβώς μεταφερόμενα θα πρέπει κάπως να αναγνωρίζεται ε, ο ενδιαφερόμενος και ε, ότι η ιδιότητά του ε, να έχουν κάρτα αναπήρου και να μπορούν να το χρησιμοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χαίρουν το δικαιωμάτων τους. Σε διάφορα κράτη-μέλη. Αυτό δεν έχει να κάνει με ποσά. Κάποιος που έχει αναπηρία στην Ισπανία την ίδια αναπηρία θα έχει αν είναι Πολωνός ή Ιταλός. Και τελικά αυτό δεν οδηγεί σε διακρίσεις. Μπορεί κάποιος να έχει κάρτα αναπήρου ισπανική και να ταξιδεύει εκτός της Ισπανίας, αλλά η ίδια αναπηρία να μην αναγνωρίζεται στη χώρα στην οποία μεταβαίνει ο, ο ανάπηρος που έχει την ισπανική κάρτα. Ταυτότητα ουσιαστικά. Επίσης, θέλουμε να ακούσουμε και τις ενώσεις εκπροσώπων ατόμων με αναπηρία. Και τέλος, ε, στο θέμα της υγείας, η έκθεση εφαρμογή για την οδηγία για ε, τη διασυνοριακή περίθαλψη ε, είχε αποτέλεσμα πάρα πολύ απογοητευτικό. Υπάρχουν διατάξεις που τιμωρούν διάφορα κράτη-μέλη. Ε, γιατί τα κράτη, εκτός του ότι αργούν να τα μεταφέρουν αυτά στην εθνική νομοθεσία, δεν τα εφαρμόζουν και βάζουν εμπόδια για να μην μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν χρήση. Ανεξαρτήτως χώρας, θα πρέπει ο Ευρωπαίος πολίτης να χαίρει γενονομική περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πολλές φορές είναι τέτοια τα εμπόδια και τέτοιοι φραγμοί που απογοητεύεται. Το άρθρο 7 θα πρέπει να εφαρμόζεται με το σωστό τρόπο, να αρθούν τα εμπόδια και οι φραγμοί που ορθώνουν τα κράτη-μέλη και να εναρμονιστεί το προπετούμενο για να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση και να, κάνει, να σκέφτεται το δικαίωμά του. Και επίσης ζητούμε εναρμόνιση των διαφόρων κριτηρίων έτσι ώστε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να έχεις και μια ευρωπαϊκή κάρτα υγείας. Και εκεί να δείτε διαφορές που έχουν τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Είναι πάρα πολύ διαφορετική η κατάσταση που επικρατεί σε κράτο μέλο. Εμείς ζητούμε να εναρμονιστούν τα κριτήρια ανεξαρτήτως χώρας. Αυτά ουσιαστικά ε, στη γνωμοδότησή μας τα βασικότερα σημεία. Thank you very much. be happy to... Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με πολύ μεγάλη χαρά να δώσω το λόγο στους ε, συναδέλφους, ε, στους Σκιώδης. Ε, κύριε Μαριά, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Μαριά, να μιλήσετε. Νομίζω έχει ζητήσει το λόγο ο Πίτερ. Θα μιλήσω μετά. Yeah. Peter for the floor, but I would like to take the coordinators first. Ε, ναι. Σιγά σιγά κουράσκα κι εγώ. Ε, ποιοι θα μιλήσουν πρώτα, οι Σκιώδης. Λοιπόν, ε, εσείς παρακαλώ. Θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η γνωμοδότηση και οι απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν από την ε, συνάδελφο. Υπάρχουν δύο-τρία επίπεδα που πρέπει να δούμε τα θέματα. Πρώτα απ' όλα στα δικαιώματα των ε, αναπήρων. Νομίζω ότι πρέπει να εμπίνουμε σε αυτό που λέμε πάντοτε σε αυτή την Επιτροπή, στην στήριξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβάλλει προς αυτή την ε, κατεύθυνση. Ταυτόχρονα πρέπει να περάσει και ένα μήνυμα προς τα κράτη-μέλη, διότι πολλά κράτη-μέλη περιορίζουν τα δικαιώματα και τα επιδόματα αναπηρίας ε, έχουμε πρόσφατα φαινόμενα στην Ελλάδα η οποία πιεζόμενη από την Τρόικα περιορίζει συνεχώς τα δικαιώματα αναπηρίας. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τις συντάξεις. Ε, υποτίθεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα στο θέμα των συντάξεων και μπορεί να παρεμβαίνει μόνο συντονιστικά. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι η Τρόικα έχει επιβάλει ιδίως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες μείωση των συντάξεων. Οι συντάξει στην Ελλάδα πλέον έχουν μειωθεί 60 με 65%. Και ενώ η Κομισιόν και γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει δεν έχει αρμοδιότητα στα θέματα των συντάξεων, στην Ελλάδα, εάν δεν μειωθούν οι συντάξει, αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να συνεχιστούν οι διαδικασίε δανειοδότηση τη χώρα. Και στην πράξη γίνεται ένα εκβιασμό. Ή μειωνεται τι συντάξει ή δεν παίρνετε την επόμενη δόση του δανείου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει πέραν των παρατηρήσεων οι οποίες έχουν τεθεί να υπάρξει και μια ειδική μνήμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως μέσω της Τρόικας στην Ελλάδα παρανόμως παρεμβαίνει και μειώνει συνεχώς τις συντάξεις. Αυτό είναι βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Οπωσδήποτε όμως τα θέματα της μεταβίβασης των δικαιωμάτων των συνταξιοδοτικών είναι σημαντικά. Όταν έχεις συνταξιοδοτικά δικαιώματα αποκτήσει σε μια χώρα, προφανώς πρέπει να έχεις δικαιώματα να τα μεταφέρεις σε άλλη χώρα. Και αυτή η διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να είναι μια διαδικασία που να μπορεί να διευκολύνεται. Το τρίτο θέμα είναι τα επιδόματα ανεργίας. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε υπέρ της δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού επιδόματος ανεργίας. Και τα δικαιώματα που αποκτά κανείς σε μια χώρα, αν είναι εγγεγραμμένος για να πάρει επίδομα ανεργίας να μπορεί αυτά να τα μεταβιβάζει σε άλλη χώρα όταν πάει να δουλέψει εκεί. Έχουμε μια τεράστια κινητικότητα. Από την Ελλάδα έχουν φύγει 500.000 νέοι για ε, να βρουν δουλειά σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιώματα τα οποία έχουν στην Ελλάδα ακόμη και σε επίπεδο δικαιωμάτων ε, για επιδόματα ανεργίας θα πρέπει να μπορούν να τα λαμβάνουν. Και κυρίως τα, επιδόματα ανεργίας πρέπει να τα λαμβάνουν όλοι οι άνεργοι. Στην Ελλάδα μόνο ένα 15% των ανέργων λαμβάνει τα επιδόματα ανεργίας. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ε, πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση η γνωμοδότηση. Θα κάνουμε και άλλες παρατηρήσεις. Αυτές ήταν οι σκέψεις οι δικές μας ως CCR ε, για την ε, γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Peter, Peter, Sie haben das Wort. Εγώ μιλώ εκ μέρους ε, του κύριου Βαλέζα που δυστυχώς ε, δεν είναι παρόν. Ε, ευχαριστεί ο κύριος Βαλέζα την εισηγήτρια Πράγματι, το θέμα πρέπει να λυθεί, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ περίπλοκο. Υπάρχουν ε, πολλές διατάξεις, ε, ε, αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους συγκεκριμένες εθνικές συνθήκες. Εδώ λοιπόν αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή των διατάξεων, δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια όπως επίσης δεν υπάρχει και σιγουριά τουλάχιστον όσον αφορά τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όπου στην νομολογία αυτή αναφέρονται πάρα πολύ σημαντικοί κανόνες ε, για τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Η πρόταση αυτή υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο τα δικαιώματα της κοινωνικής ασφάλισης ε, να μπορεί κανείς να τα προστατεύσει. Ε, το σημαντικότερο τμήμα της πρότασης αφορά την πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα τα οποία προσφέρονται σε ανέργους, σε, ε, περίπτωση ε, άδεια μητρότητα, ε, ανεργίας υπάρχουν οικογενειακά επιδόματα τα οποία θα πρέπει να χορηγούνται ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν ειδικέ ρυθμίσει από αυτόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει πάρα πολλέ αναφορέ που ακριβώ εξετάζουν το θέμα του συντονισμού των διαφόρων επιδομάτων ε, την δυνατότητα του να χορηγούνται επιδόματα σε περίπτωση παραδείγματο χάρη ασθενεία. Ο κύριο Βαλέντσα υπογραμμίζει ότι αυτό το θέμα είναι πολύ μεγάλη σημασία και χαίρεται ήδη για την αγαστή συνεργασία με την κυρία Κάμπερσον, του και ηγητέ. Ε, αυτά είχαμε να σα πούμε για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Mrs. Kuneva, try to be very short. We are losing tempo. Κυρία Κούνεβα, αν έχετε καλοσύνη σύντομα, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, βουλευτέ, παίρνω το λόγο ω καλεσθήτρια τη Γκουέντζα για το σχέδιο γνωμοδότηση που αφορά τι αλλαγέ του κανονισμού για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση. Το σχέδιο συνέταξε την Επιτροπή Αναφορών η Σολεντάτ Ρουίτ και την οποία ευχαριστώ. Την ευχαριστώ γιατί πολύ σωστά στην έκθεση τη, εστίαζε και ενέδειξε τους ανθρώπους με αναπηρίες καθώς και τους σπουδαστές. Δηλαδή έφερε στην επιφάνεια αυτές τις δύο μεγάλες κοινωνικές ομάδες τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αγνοεί ότι παρουσιάζουν κινητικότητα και έχουν τα ίδια δικαιώματα σε μεταφορά των δικαιωμάτων τους όταν αλλάζουν χώρα διαμονής και εργασίας. Κάποιοι μπορούν να πούν, μα παρουσιάζουν και τα άτομα με αναπηρία κινητικότητα φυσικά. Οι υποφαινόμενοι, για παράδειγμα, έφυγα από τη Βουλγαρία και βρέθηκα να εργάζομαι στην Ελλάδα. Και από εκεί με βαριά αναπηρία, πολύ πριν από την εκλογή μου, μετακινήθηκα στην Γαλλία. Όσοι από τους σπουδαστές και τα δικαιώματα τους, στα οποία σωστά επικεντρώνει η συγκίτρια, αν και φαίνεται να ξεχνάει η Κομισιόν, δεν χρειάζεται να πω πολλά Έχουμε πια μια γενιά που για να εξασφαλιστεί πτυχία, υψηλή εξειδικευσή, κατάρτιση και δεξιότητε, μετακινείται με ευκολία από χώρα σε χώρα. Μεγάλο το θέμα της ενδοευρωπαϊκή κινητικότητα, που είναι ουσιαστικά μια μετανάστευση από το ένα κράτος μέλος σε άλλο και φυσικά δεν αφορά μόνο τις χώρες της Ανατολική Ευρώπη, Αφορά όλο το Ευρωπαϊκό Νότο. Ιδού τα τελευταία στοιχεία που έδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον αριθμό των ανθρώπων που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Από το 2010 μετανάστευσαν 700.000 άνθρωποι. Ο ρυθμός των εισερχόμενων μεταναστών από το 40.000 του χρόνου μέχρι το 2009 ανέβηκε στις 109.000 και συνεχίζει να, αυξάνεται. Βασικοί ευρωπαϊκοί προορισμοί η Γερμανία, η Βρετανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Θεωρώ πολύ σωστέ και προτείνω να υποστηριχτούν οι τροπολογίε 1 έως 7 γιατί προβάλλουν την ανάγκη να προωθηθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρία και να διασυνδεθεί τόσο με την Ευρωπαϊκή Κάρτα κοινωνική Ασφάλιση, που και αυτή δεν υπάρχει και πρέπει να δημιουργηθεί όσο και με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλιση ασθενείας που υπάρχει. Επίση, συμφωνώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσει κατά των ανθρώπων που δεν αναζητούν εργασία. Γιατί δεν πρέπει μόνο ο κάθε εργαζόμενος να έχει κοινωνική προστασία, αλλά ο κάθε άνθρωπος που και αν βρίσκεται, όπου και αν βρίσκεται. Συμφωνούμε και με τις τροπολογίες 1 και 2 που θέτουν ζητήματα κοινού ορισμού και κριτήρια για την αναπηρία. Αλλά τα επιμείνουμε ώστε οι παροχές μακροχρόνιας φροντίδας να μην ενταχτούν σε ξεχωριστό κεφάλαιο, αλλά να προσθετούν στο κεφάλαιο για την ασφάλιση της ασθένειας, ώστε κανεί, κανείς δικαιούχος να μην αποκλειστεί από αυτέ. Σε αυτό το σημείο θα καταθέσω τροπολογίες και ήθελα να σα ενημερώσω ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δύο χρόνια έκανε ένα πολύ μεγάλο έργο και ένταξε στην νομοθεσία τη, όλη η ρύθμιση από την ΟΗΕ για την αναπηρία για, για τους ανθρώπους με αναπηρία οριζόντια. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βάζει και κάτι παραπάνω που δεν έχει τώρα με το θέμα επευθείας αλλά σχεδιάζει να κάνει α, Ωραία, εντάξει. Αυτό που τα κάνει συνήγορο των αναπήρων, το οποίο τα βοηθήσει πάρα πολύ στους ανάπηρους να μάθουν τα δικαιώματά τους και να ξέρουν πώς να μεταχειρίζουν τη ζωή τους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά βιαζόμαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Ε, now, Έχουμε κανέναν άλλον για αυτό το θέμα? Όχι. Έχουμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολύ... Κυρία Σδάνοκα και εσείς θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Χάνετε το μικρόφωνο της ομιλητρίας. Μας συγχωρείτε, δεν ακούσαμε. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Χαίρετε και να συγχαρώ την συντάκτρια της γνωμοδότησης γιατί έχει κάνει για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει συμπεριληφθεί στην κοινή δήλωση των θεσμικών μας οργάνων για τις ε, διοργανικές προτεραιότητες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν για μας όταν ρωτά κανείς Ευρωπαίος ε, ποιο είναι το πιο σημαντικό ευρωπαϊκό αγαθό για αυτούς, συνήθως είναι το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν θα υπήρχε δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς κανόνες για συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών όταν ε, μετακομίζουν σε μια άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες δεν είναι καινούργοι υπάρχουν από το 1959 και ε, υπάρχει τακτική επικαιροποίηση ώστε να λαμβάνονται υπόψη και οι εξελίξεις των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και η πραγματικότητα φυσικά. Ε, ένα στοιχείο είναι ότι ε, οι κανόνες δεν εναρμονίζουν τα εθνικά συστήματα. Αυτό δεν είναι εθνική ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά ε, περιλαμβάνουν κανόνες για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις ε, ε, διασυνοριακά. Η πιο πρόσφατη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση είναι το Δεκέμβριο του 2016. Αυτή είναι η πρόταση που εξετάζεται σήμερα, που αντανακλά τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δίκαιη εργασιακή κινητικότητα, επικαιροποιεί τους κανόνες και προσπαθεί να εφαρμόσει σωστά ε, το συντονισμό. Είναι δίκαιη πρόταση γιατί διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία και βοηθά ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και φυσικά προσφέρει και εργαλεία στις εθνικές αρχές να καταπολεμήσουν τους κινδύνους κατάχρησης ή απάτης. Επίσης, η πρόταση ε, δημιουργεί μια πιο στενή σχέση μεταξύ του τόπου στον οποίο ε, δίνονται οι εισφορές ε, και του τόπου στον οποίο γίνεται η αίτηση για επιδόματα και δημιουργεί συγκρούσεις μεταξύ των κρατών. Ε, υπάρχουν πέντε βασικοί τομείς, η ανεργία, ε, μακροπρόθεσμα ε, επιδόματα φροντίδας, ε, επιδόματα για άτομα τα οποία είναι οικονομικά ανενεργά, κοινωνικά δικαιώματα για τους αποσπασμένους εργαζομένους και εργασιακά επιδόματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε, να διευκολύνουμε τη διαδικασία, να προχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε την Επιτροπή για την πολύτιμη συνεισφορά τη και προσβλέπουμε στη γνωμοδότησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Για μα είναι προτεραιότητα και σημαντική μάλιστα. Ευχαριστώ Σολεδά για ε, την ταχεία διεκπαιρέωση. Προθεσμία κατάσταση τροπολογιών 27 Δευτέρου στις 3 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε στις 24 Απριλίου και στην Επιτροπή Απασχόλησης στις 19 Ιουνίου. Ωραία. Γρήγορα, γρήγορα θα πρέπει να περάσουμε στο τελευταίο θέμα πριν τελειώσουμε που είναι 6 λεπτά ο χρόνος που μας απομένει. Εγώ είμαι ε, συντάκτρια της νομοδότησης για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016. Με χαρά σας παρουσιάζω το σχέδιο γνωμοδότησής μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για την Επιτροπή μας και ας ελπίσουμε ότι θα είναι ε, και χρήσιμο για την αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή που είναι η Επιτροπή ε, νομικών Θεμάτων. Ανεπαρκής καμιά φορά και κακή εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου είναι ο λόγος για τον οποίο προσφεύγουν σε εμά οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Επιτροπή Αναφορών. Η εφαρμογή ε, του Ευρωπαϊκού Δικαίου εδράζεται στις ε, συντρέχουσες αρμοδιότητες και στην κατανομή ε, αρμοδιοτήτων ε, κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από κοινού θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη και θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό γιατί εμείς από τις αναφορές που λαμβάνουμε εδώ βλέπουμε σαφέστατα στοιχεία του γεγονότος ότι ακόμα πολύ συχνά ε, μεταφέρεται ανεπαρκώς, αργά και με λάθος τρόπο η ε, νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο ε, και σε μερικές περιπτώσεις καθόλου ή δεν εφαρμόζεται σωστά. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι θεματοφύλακα των συνθήκων οφείλει να διορθώσει την κατάσταση. Αφού είναι γνωμοδότηση μπορούμε το κείμενο να το κρατήσουμε ευσύνοπτο και μικρό και να περιοριστούμε στα θέματα της δικής μας Επιτροπής. Ορίστε, σε δύο λεπτά τα είπα, προσβλέπω στις δικές σας τροπολογίες. Με χαρά σας δώσω το λόγο κύριε Μαλίνοφ. Ε, ζητώ συγγνώμη, ευχαριστώ ε, και παίρνω το λόγο για να σας συγχαρώ για το εξαιρετικό σχέδιο γνωμοδότησης ε, ήταν δύσκολη η σημερινή συνεδρίαση και εκφράζω τη συμπαράστασή μου. Ε, είναι καλό να παραμείνουμε νυφάλιοι και χωρίς πάθος στη συζητήση μας. Το θέμα είναι τεράστιο. Ε, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Εμείς θα πρέπει να το δούμε μόνο από τη δική μας σκοπιά της Επιτροπής Αναφορών. Τρεις τροπολογίες θα κάνω, να σας πω σε ποια κατεύθυνση θα πάνε. Ε, νομίζω ότι πάντα να, ε, πρέπει να τονίζουμε το βασικό ρόλο που διαδραματίζει η Επιτροπή Αναφορών πάντοτε και θα κάνω και σχετική τροπολογία. Επίσης θέλω να τονίσω την ανάγκη για μεγαλύτερη και περισσότερη διαφάνεια, ιδιαίτερα ε, στα πιλωτικά ε, προγράμματα και ε, τις προσφυγές επιβαραβάση και το διαμεσολαβητή. Και ένα τελευταίο που θέλω να τονίσω που ανησυχεί πολλούς αναφέρονται στην Επιτροπή μας και πολλές αναφορές, πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι η διαφορά της ποιότητας ε, προϊόντων τροφίμων της ίδιας μάρκας, του ίδιου εμπορικού σήματος που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μεγάλο πρόβλημα αυτό σε πολλά κράτη-μέλη και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι χάρη στις αναφορές που γίνονται και άλλα μέσα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ γρήγορα αντιδρά και με νέα μεθοδολογία που υιοθετεί. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν, αλλά καλό θα ήταν να δώσουμε ένα παράδειγμα που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως απόδειξη ότι μπορούμε να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα από τη δουλειά μας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για την καλή γνωμοδότηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά και για την ακριβία σας. Η κυρία Πρόεση. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσω θερμά ε, για αυτό το πολύ καλό σχέδιο. Τα περισσότερα σημεία της ε, γνωμοδότησης ε, τα υποστηρίζω. Προφανώς και είναι σωστό στους πολίτες να παρουσιάζουμε μια θετική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποτεδήποτε υπάρχουν δυσάρεστες καταστάσεις θα πρέπει και αυτές να αναφέρονται. Εγώ θέλω να πω ότι παρόλα αυτά πολλά πράγματα δεν εξετάζονται όπως πρέπει. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αναφορών με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Κυρίως ε, αναφορές ε, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε οδηγία επί παραβάση. Σε αυτή τη γνωμοδότηση νομίζω ότι είναι σημαντικά, σημαντική όλη η νομική τομή σε πιο συγκεκριμένα για το 2016 πρόκειται για την κοινή αγορά, τη δικαιοσύνη και για το περιβάλλον. Οι δικές μου οι τροπολογίες ε, θα ε, ασχοληθούν ακριβώς με αυτά τα θέματα. Και χαίρομαι που ε, αναφέρεστε σε μια μεταναστευτική πολιτική, πολιτική τρομοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα αυτά θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δυστυχώς βέβαια εξακολουθεί να μην υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε, να δούμε πώς ακριβώς τα κράτη-μέλη εκπληρούν τις υποχρώσεις τους. Χαίρομαι για τη συνεργασία μαζί σας και με άλλους εισηγητές, με τους οποίους ε, θέλουμε να συμβάλλουμε έτσι ώστε να έχουμε καλύτερη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μαριάς. Λοιπόν, για να δούμε αν θα τα καταφέρετε σε 30 δευτερόλεπτα. Να σας ευχαριστήσω κυρία Πρόεδρε για την ε, ε, γνωμοδότηση αυτή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κάνουμε τις παρατηρήσεις μας βεβαίως και με τις τροπολογίες. Θεωρώ πιο σημαντικό το θέμα της εφαρμογής του ελέγχου μάλλον της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος που παίζει η Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ σημαντικός και θεωρώ επίσης ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να επιδείξουν αλληλεγγύη στα θέματα των προσφύγων. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και η Ιταλία δεν αντέχουν άλλους πρόσφυγες πλέον και παράνομους μετανάστες και θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει ποιες χώρες δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις αλληλεγγύης για να τις καλέσει να συμμορφωθούν προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε λοιπόν τι να κάνουμε τώρα. Now the floor is to the Commission, Mr. Slotjes. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. I'm sorry. Συγγνώμη, ο κύριο Σόλτες. Α, περίπου, μοιάζουν τα ονόματά σας που βλέπω εδώ γραμμένα και νομίζω ότι ήταν εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. δεύτερα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο για τη γνωμοδότηση αυτή. Δεύτερον, συμφωνώ ότι η σωστή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκ των όνου κάνευ για όλους τους Ευρωπαίους. Και επίση τρίτον, χαιρετίζω τη δυνατότητα των Ευρωπαίων πολιτών να στέλνουν ε, αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά αν μου επιτρέπει και κάποιες προτάσεις να κάνω. Θα κάνουμε κάποιες τροπολογίες στο κείμενό σας, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να εκφράσουμε και κάποια μικρή κριτική ε, ως προς την εφαρμογή του δικαίου. Από την άλλη εβδομάδα θα σας κάνουμε τις τροπολογίες για να βελτιώσουμε λίγο το κείμενο. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ και περιμένω τη συνεισφορά σας, προφανώς, αλίμονο για να βελτιώσουμε περαιτέρω το κείμενο και να το κάνουμε και πιο ενδιαφέρον και ελπίζω για να μας λάβουν πιο ε, σοβαρά υπόψη. Τώρα ο κύριος Σλότσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μοιάζουν τα ονόματα που λέμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης. Καλωσορίζουμε τις ε, συστάσεις σας. μα ε, βοηθούν πάρα πολύ και τις προτάσεις σας. Σημειώνουμε που θέλετε να δείτε βελτιώσεις και ως προς τη διαφάνεια και στην αιτήσια έκθεση. Δίνουμε ε, παραδείγματα πραγματικά όπου οι αναφορές κάνουν τη διαφορά. Ε, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για τον αριθμό τους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ότι χρειάζεται ενημέρωση, τα δεδομένα και η αντίστοιχη μηχανοργάνωση που πάντα δεν έχουμε ε, τη δυνατότητα. Πολλές φορές ο κόσμος κάνει ταυτόχρονα και αναφορές και καταγγελίες. Ε, υπάρχει κάποια σύγχυση ως προς τους αριθμούς. Εκφράζεται μια ανησυχία για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τη δυνατότητα να παραπέμπουμε τους αναφέροντες και τους καταγγέλλοντες σε άλλους μηχανισμούς ε, ε, διόρθωσης ή συμμόρφωσης όταν είναι περιορισμένη η δυνατότητά μας. Εμεί δεν του εγκαταλείπουμε στη μοίρα του, αλλά δεν υπάρχει πάντα δυνατότητα προσφυγή σε άλλο οργανισμό. Αν υπάρχει κάποιος ε, επιτόπιος μηχανισμός που μπορεί να τους βοηθήσει καλύτερα, ε, τους συμβουλεύουμε γιατί μπορεί να κινδυνεύσουν να απογοητευτούν όταν αρχίσει μια ολόκληρη διαδικασία προσφυγής επί παραβάση που παίρνει πάρα πολύ χρόνο και μπορεί τελικά να μην δικαιωθούν. Ε, σταματώ εδώ γιατί δεν υπάρχει και χρόνος. Και πεινάμε και τρέχουμε όλοι για φαγητό, λέει η Πρόεδρος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων που αυξάνεται και εντείνεται και γίνεται όλο και πιο καλή. Ευχαριστώ πολύ και να χαρείτε τον ήλιο.